Okay, ladies and gentlemen, we continue our session. Wie wir besprochen Κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Όπως είπαμε, έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει η σειρά των θεμάτων ε, στην ημερήσια διάταξη. Ε, θα ασχοληθούμε Πρώτα με την μεταρρύθμιση των κανόνων περικρατικών ενισχύσεων στι υπηρεσίε ε, κοινή ωφελία. Χωρί πολλά πολλά, να δώσω το λόγο στον ε, συνάδελφο Χέκμαρκ, που είναι ο εισηγητή ε, για το θέμα αυτό από την Επιτροπή μα. να έχει το λόγο. Εκτός μικροφώνου δεν ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Το βασικό μου μήνυμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στις κρατικής ενισχύσεις και τις ενισχύσεις που κάνουν τις υπηρεσίες αυτές πιο προσβάσιμες στον απλό πολίτη. Είναι σημαντική η διαφορά αυτή, διότι συνήθως αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να διασφαλίσουμε οι πολίτες μας να λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Και γνωρίζουμε ότι όσο πιο, σημαντικό, όσο πιο σημαντικές είναι οι υπηρεσίες, τόσο πιο σημαντικό είναι να είναι υψηλής ποιότητας. Και πάντα θα πρέπει να στηρίζουμε την ανάπτυξη πιο ε, οικονομικών ε, και πιο αποτελεσματικών ε, υπηρεσιών και τα μονοπόλια πάντα εμποδίζουν κάτι τέτοιο. Όσο περισσότερο λοιπόν μπορούμε να ανοίξουμε την εσωτερική αγορά για τις υπηρεσίες που σήμερα περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες κοινή ωφελία, τόσο καλύτερο είναι, διότι τόσο πιο ευρεία θα είναι η επιλογή για τον κάθε πολίτη. Θα ήθελα όμως να σας θυμίσω τις ε, εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Για πολύ καιρό σε όλες τις χώρες μας υπήρχε μονοπόλιο στον τομέα αυτό με πολύ μικρή ανάπτυξη των υπηρεσιών αλλά και πολύ μικρή ανάπτυξη όσον αφορά το, τη μείωση του κόστους και την ε, αποτελεσματικότητα. Τώρα που απελευθερώθηκε αυτός ο τομέας της οικονομίας είδαμε ε, μεγάλες επιχειρήσεις ε, στα πλαίσια μιας δυναμικής οικονομίας και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε το ίδιο και σε μια σειρά άλλων τομέων όσον αφορά τις υπηρεσίες ε, κοινή ωφελία. Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα κατά της δυνατότητας του πολίτη να έχει επιλογές. Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα εάν μας ενδιαφέρει ο μεμονωμένος καταναλωτής διότι θα έχει καλύτερες υπηρεσίες από ό,τι πριν. Σε διάφορες χώρες, στα διάφορα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις σχετικά με την χρηματοδότηση των υπηρεσιών αυτών. Και ο βασικός μου στόχος ε, με αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης είναι να φροντίσω να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται τις ε, ευκαιρίες αυτές ε, στο μέλλον τους τομείς αυτούς, ε, επιτρέποντας τους τομείς αυτούς να αναπτυχθούν, ε, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το συμφέρον ε, του κάθε πολίτη. Προσλέπω λοιπόν στην συζήτηση και στις τροποποιήσεις που θα λάβω. Θα κλείσω εδώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ θερμά. Πρώτα να δώσω το λόγο στην κυρία Τζαβέλα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Χόκμαρκ για το λακωνικό και πολύ περιεκτικό κείμενό και για τις ε, φωτισμένες και προς το μέλλον προτάσεις του. Ε, θα ήθελα να προτείνω μία ε, τροπολογία ή μία προστίκη, όχι τροπολογία, μία προστίκη στην παράγραφο 3, κύριε Πρόεδρε. Επειδή έχω την εμπειρία από το Broadband Report που ήμουνα εισηγήτρια όταν διάβασα τους κανόνες του State Aid για το broadband ήταν πάρα πολύ πολύπλοκες. Γι' αυτό η τροπολογία την οποία θα πρότεινα στην παράγραφο 3 είναι να προσθέταμε στην πρώτη πρόταση affordable prices for citizens and simplification of the rules και απλοποίηση των κανόνων. Αυτή είναι η, η προσθήκη την οποία θα πρότεινα κύριε Χόκμαρκ ε, στο κείμενό σας γιατί θα πρέπει να είναι κατανοητοί και απλοί οι κανόνες για να γίνονται και εφαρμοστέοι από όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάμπερτς. Δεν ε, είμαστε πολλοί παρόντες. Ήθελα να ε, εκφράσω κάποιες γενικές ε, σκέψεις. Ο κύριος Χακμαρή είναι από τους πιο φιλελεύθερους από όλη την ομάδα του ΕΛΚ και είσαστε πιστό στην παράδοσή σας. Εγώ ήθελα να πω το εξή. Συμμερίζομαι δύο θέσεις. Πρώτον, ότι γενικά οι κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να είναι οικονομική φορής ε, με την βασική έννοια του όρου. Οι εποχές που οι κυβερνήσεις ήταν ε, οι οικονομικοί φορεί που είχαν ξενοδοχεία, που ήταν παραγωγή αυτοκίνη, κατασκευαστέ αυτοκινήτων κλπ. Έχουν περάσει οι εποχέ αυτέ. Δεύτερον, συμμεριζόμαστε τη θέση ότι οι ε, πολίτες ε, θα πρέπει να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Ωστόσο, ε, θα διαφωνήσω μαζί σας στο ότι η μεταβίβαση περισσότερων δραστηριοτήτων από τον ε, δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα ε, θα οδηγήσει σε καλύτερες υπηρεσίες ή χαμηλότερες τιμές. Ε, εδώ θα διαφωνήσω και αν κοιτάξουμε τις τηλεπικοινωνίες που αναφέρετε εσείς στο σχέδιο γνωμοδότησής σας, διαπιστώνουμε ότι ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας, της οποίας στηρίξαμε την ε, ιδιωτικοποίηση στις χώρες, ιδιαίτερα στις χώρες όπου ήμασταν ε, στην εξουσία όταν έγινε αυτό. Αυτό που διαπιστώσαμε εκ των υστέρων είναι ότι αυτοί που επωφελήθηκαν από, αυτές τις, ε, από αυτή την απελευθέρωση είναι οι πελάτες επιχειρήσεις. Οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν όχι για τους καταναλωτές, η ιδιωτικοποίηση ε, έκανε το κρατικό μονοπόλιο, η ιδιωτικό ολιγοπόλιο. Ε, γενικά όμως καταλήγουμε σε ολιγοπόλιο, δεν καταλήγουμε σε ελεύθερη αγορά. Αν κοιτάξουμε την ε, προμήθεια ενέργειας στη Γερμανία, υπάρχουν τρεις ή τέσσερις προμηθευτές. Ε, στη δική μου χώρα, σε τούτη τη χώρα που βρισκόμαστε, υπάρχουν ε, αρκετέ επιχειρήσει, αλλά η μία κατέχει το 85% τη αγορά. Με την ιδιωτικοποίηση, λοιπόν, δεν είδαμε αμέσω ε, πλεονεκτήματα στην αγορά και αυτήν την παρατήρηση ήθελα να κάνω. Γενικά, το ύφο του κειμένου υπονοεί ότι αν ακολουθήσουμε την κατεύθυνση αυτή θα έχουμε όλα τα ωφέλη. Δεν λέω ότι το αντίθετο ισχύει, αλλά ε, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί ε, όσον αφορά τις διατυπώσεις που λένε ότι αν ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση θα έχουμε ε, ωφέλη για όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες αποχρώσεις στο κείμενο. Θα προσπαθήσουμε να σας υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ λογικά και φρόνιμα ήταν όπως πάντα τα λόγια του εισηγητού και πολύ σωστά ε, ξεχώρισε με σαφήνεια τους τομείς τους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Και όπως είπατε δίνουμε τη βοήθεια για να βοηθήσουμε τους καταναλωτές, τους πολίτες και όχι κατά ανάγκη τις ε, εταιρείε. Πολύ σωστά το διευκρινίσατε. Και στις τηλεπικοινωνίες έχουμε δει μια πραγματική επανάσταση που έχει εξασφαλίσει καλύτερες υπηρεσίες για ε, ένα τεράστιο αριθμό του πληθυσμού. Αλλά υπάρχουν θύλακες ε, και ε, για κάποιους πολίτες είναι απρόσιτες ακόμη αυτές οι υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιοχές της Αγγλίας δεν έχουμε καν σήμα κινητού, για να μην μιλήσω για ευρυζωνία. Οπότε αυτή η θύλακες, η δυσπρόσιτη, είναι το πρόβλημα για κάθε κλάδο και εκεί θα πρέπει να ε, ενισχύσει το κράτος προσφέροντας τη βοήθεια. Και αυτούς τους δύσκολους καιρούς ε, που θέλουμε επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες στις, ε, και στην ενέργεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με πιο ορθολογικό τρόπο και τα δημόσια και τα ιδιωτικά κονδύλια. Γιατί θα πρέπει τα δημόσια κονδύλια να δώσουν μόχλευση για τα ιδιωτικά θα φροντίσουμε με τις τροπολογίες μας όχι να διευκρινίσουμε τους κανόνες αλλά να ε, επιταχύνουμε την διευκρινίσή τους γιατί πολύ συχνά ε, ορισμένα καλά σχέδια προσκρούν σε εμπόδια επειδή είναι μικρής εμβέλειας και επειδή δεν υπάρχει σαφήνεια σε ό,τι αφορά την ε, παραβίαση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, το σχέδιο κολλάει και πολλοί φοβούνται και δεν ζητούν διευκρινήσεις ε, για να μην προσκρούσουν σε αυτούς τους κανόνες ε, για την απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων. Σωστό λοιπόν είναι να γίνει αυτή η διευκρίνηση εγκαίρως ώστε να βοηθήσουμε τη σύμπραξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για επενδύσεις. Η κυρία Μαντουρέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κύριου Γκάλφιν, του σκιώδου συγγητού μας, που δεν μπόρεσε να έρθει, βρίσκεται στην πατρίδα του και με επιφόρτησε να σας διαβιβάσω κάποιες παρατηρήσεις, ε, κυρίως να τις διαβιβάσω στον εισηγητή της γνωμοδότησης, τον κύριο Χέκμαρκ. Φυσικά τον ευχαριστεί για την προσπάθειά του και το εγγραφό του, αλλά έχει τη γνώμη ότι ίσως αυτή η γνωμοδότηση δεν στηρίζει αρκετά τη θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Φαίνεται ότι στόχο έχει να βοηθήσει τις μεγάλες επιχειρήσεις αυτή η γνωμοδότηση. Αυτή είναι η γνώμη του Σκιώδου Σιγητού. Βέβαια αυτό είναι συζητήσιμο. Θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε και άλλα σημεία που να ενισχύει πραγματικά τη θέση και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μου λέει λοιπόν ο Σκιώδης Ηγητής ότι στο πρώτο σημείο δεν μιλούμε για τη μείωση των ορίων ε, των δημοσίων προμηθειών, κάτι που θα ήταν πολύ σημαντικό για την απλούστευση. Μου είπε ότι συμφωνούμε με το 2.5, αλλά κατά τη γνώμη του είναι ανεπαρκής η διατύπωση και θα πρέπει να την ενισχύσουμε. Δεύτερη παρατήρηση του σκιώδου είναι σημαντικό να προσθέσουμε και το θέμα της καινοτομίας που απουσιάζει αυτή τη στιγμή από το κείμενο και επίσης συμφωνεί και ο δισηγητής με την πρόταση ε, να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διευκολύνει ε, την ε, διαφανή, απλούστερη και πιο προσιτή χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να εξασφαλίσουμε απρόσκοπτη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις κρατικές ενισχύσεις. Αυτά ήταν συντομία τα σχόλια εκ μέρους του σκιώδου συζητήτου μας. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ε, η Κομισιόν θέλει κάτι να πει, ίσως δεν είναι απαραίτητο, τότε θα πρότεινα το εξής. Είχαμε την τροποποίηση αυτή στη μερισσία διάταξη. Συμφωνήσαμε να προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα το θέμα αυτό. 11 ε, Σεπτεμβρίου η ε, υποβολή τροπολογιών ε, και μάλιστα στα αγγλικά έτσι συμφωνήσαμε. Ωραία. Ο συνάδελφος Χεκμαρκ... Θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στον συνάδελφο Χεκμαρκ. Ε, ναι, επιτρέψτε μου να απαντήσω σύντομα σε κάποιες από τις παρατηρήσεις. Καταρχήν, να απαντήσω λίγο ρητορικά, απευθυνόμενο σε κανέναν αλλά σε όλους ε, και ίσως ιδιαίτερα στον Φίλιπ. Μερικέ φορέ με απασχολεί ότι όταν μιλάμε για τις καλύτερε δυνατές ευκαιρίε για τους καταναλωτέ. αυτό θεωρείται φιλελευθερισμό ή κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν συμφέρον και των πρασίνων. Ε, θέλετε κάτι άλλο από το ε, καλύτερο συμφέρον του καταναλωτή. Ή μερικές φορές λέγεται ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα στο παρελθόν. Πότε δεν συμφωνώ με ανθρώπους που λένε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα στο παρελθόν. Όταν κάποιο μου λέει ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα στο παρελθόν, εγώ λέω ότι όχι, αυτό δεν ισχύει. Εσεί ήσασταν ίσω καλύτερο στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι όταν εξετάζουμε μια σειρά σημαντικών ε, υπηρεσιών κοινή ωφελία, βρίσκονται στον πυρήνα του οικονομικού μας μέλλοντος και θα πρέπει να κάνουμε την επιλογή. Θέλουμε ανάπτυξη πλουραλισμό στην παροχή των υπηρεσιών ή όχι. Αν θεωρείτε ότι αυτή είναι ριζική απάντηση, νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να ανησυχήσουμε, διότι πότε-πότε πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, να στηριζόμαστε σε αυτά που έχουμε σήμερα. Και η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση. Και θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Μήπως δεν κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Μήπως μπορούμε να έχουμε δυναμική ανάπτυξη σε μια σειρά τομέων, όπως είδαμε άλλωστε και στις τηλεπικοινωνίες. Ε, νομίζω ότι και εσείς και εγώ και όλοι συμφωνούμε. Συμφωνώ ε, ότι σε κάποιες χώρες ο τρόπος που έγινε η ιδιωτικοποίηση δεν ήταν ε, ο καλύτερος δυνατός. Γι' αυτό πιστεύω ότι κρίσιμο είναι να υποστηρίξουμε τους πελάτες, τους καταναλωτές. Και αν πιστεύετε ότι αυτή είναι ριζική λύση, ε, τι να σας πω, επασεπτώσει, να, να σταματήσω να είμαι κακός, θα ήθελα να... Ε, ε, σας καλέσω να υποβάλλετε τροπολογίες όσον αφορά αυτό που υπόθηκε για την απλοποίηση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε πιο ξεκάθαρους κανόνες. Η απλοποίηση δεν σημαίνει μόνο πιο εύκολους ε, κανόνες, ε, σημαίνει και πιο ε, εύκολους στην εφαρμογή τους κανόνες. Όσο περισσότερους κανόνες έχουμε, όσο πιο πολύπλοκα είναι τα πράγματα, τόσο πιο δύσκολα είναι. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Και επίσης, όπως τόνισε η κυρία Τζαβέλα, είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα για πιο γρήγορη λήψη αποφάσεων. Όταν έχουμε συζήτηση σχετικά με το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες ε, στην Ευρώπη, μην λέτε ότι αυτά είναι ριζοσπαστικά πράγματα, γιατί αν αυτά είναι ριζοσπαστικά τότε βρισκόμαστε ε, σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν νομίζω ότι χρησιμοποίησα ποτέ τη λέξη ριζοσπαστικός, ε, απαντάει ο κύριος Λάμπερτς. Ωραία. Έτσι ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε συμφωνήσει σχετικά με τις ε, προθεσμίες. Ε, σας ευχαριστώ θερμά και μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, το σημείο 5 προς την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας μέχρι το 2014. Να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Ένα λεπτό, να περιμένουμε ένα λεπτό να προσέλθει στο βήμα εκπρόσωπο της Κομισιόν. begrüße ganz herzlich Frau Bernhards, Head of Καλωσορίζω θερμά την κυρία Μπένα που, που είναι επικεφαλή ε, της ε, μονάδας για το ηλεκτρικό ρεύμα και το αέριο της Κομισιόν. Θα μιλήσουμε για την έκθεση σχετικά με την κατάσταση της αγοράς ενέργειας. Θα θυμάστε ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2011 Ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε το στόχο μέχρι το 2014 να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ε, ενέργεια Στο μεταξύ έχουν γίνει πολλά. Είδαμε τα ότι ε, ως συμπέρασμα από τα γεγονότα της Φουκουσίμα πολλές χώρες έχουν αποφασίσει να τροποποιήσουν την πολιτική ενέργειά τους. Ε, όταν όμως ε, χώρες λαμβάνουν αποφάσεις ε, μόνες τους, τότε αυτό αντίκειται στην εσωτερική αγορά. Και έτσι δεν κινούμαστε προς την κατεύθυνση μιας εσωτερικής αγοράς, αλλά προς την κατεύθυνση πιο ισχυρών εθνικών πολιτικών ενέργειας. Γι' αυτό χαίρομαι που βρίσκεται εδώ σήμερα εκπρόσωπος της Κομισιόν για να μας παρουσιάσει την κατάσταση των την κατάσταση του ενεργειακού τομέα. Κυρία Μπέναρτ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να είμαι μαζί σας σήμερα και να σας παρουσιάσω από πλευράς της Επιτροπής την κατάσταση ολοκλήρωσης της αγοράς ενέργειας για το 2014 και να σας δώσω επίσης στοιχεία για το που βλέπουμε εμείς τα βασικά προβλήματα στο μέλλον και να ακούσω και τους συναδέλφους σας και τις αντιδράσεις σας και ίσως να απαντήσω και σε κάποιες πιθανώς ερωτήσεις που θα θελήσετε να θέσετε. Η ολοκλήρωση της ε, εσωτερικής αγοράς ενέργειας είναι στόχος πάντα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το είπαμε και στο τελευταίο Συμβούλιο Ενέργειας. Το θέμα δεν είναι να αντιμετωπίσουμε μόνο το θέμα της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στα πλαίσια της Ευρώπης 2020, αλλά και τα θέματα διασφάλειας προμήθειας ενέργειας, κλιματολογικών αλλαγών και ένταξης των ανανεώσιμων πηγών. Όταν μιλάμε για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μέχρι το 2014, τι ακριβώς εννοούμε. δύο βασικές διαστάσεις. Καταρχάς, το ποσοστό ανοίγματο της αγοράς στην ανταγωνιστικότητα. Το δεύτερο στοιχείο, εξίσου σημαντικό με το πρώτο, είναι το θέμα της ολοκλήρωσης της αγοράς αυτής. Ιστορικά, οι αγορές της ενέργειας, περισσότερο από άλλες αγορές όπως των τηλεπικοινωνιών, έχουν εθνικές διαστάσεις με εθνικούς σχεδιασμούς και αρχιτεκτονικές. Είναι δύσκολο λοιπόν να τα συνδυάσουμε αυτά και να υποφεληθούμε από μια ενιαία αγορά. Ο πρόεδρος Ρόιλ ζήτησε να μάθει πού βρισκόμαστε σήμερα και αν πράγματι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη. Αν δει κανεί την πρώτη διάσταση, το άνοιγμα των αγορών, Υπόθηκε ήδη ότι πράγματι βλέπουμε αρκετούς που εμπλέκονται στην αγορά αυτή, αυξάνεται ο αριθμός αυτών που εμπλέκονται στις διάφορες αγορές ενέργειας στα κράτη-μέλη. Κάποιες χώρες που παλιά είχαν στον εθνικό χώρο τους έναν να τώρα στις περισσότερες βλέπει κανείς ότι υπάρχουν πολλαπλοί πρωταγωνιστές για το εάν αυτό οδηγεί πράγματι σε μια δυναμική κατάσταση του ανταγωνισμού στο λιανικό εμπόριο ενέργειας αυτό είναι διαφορετικό. Γιατί είναι αλήθεια ότι θα πρέπει μερικές φορές να αντιμετωπίσουν ένα παραδοσιακό παροχέα. Στο Βέλγιο, σαν παράδειγμα, στον ηλεκτρισμό βλέπει κανείς ότι σε επίπεδο παραγωγής ελέγχεται από έναν παροχέα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και το ίδιο ισχύει και στη Γαλλία κτλ. Η δυναμική την οποία παρέχει ο ανταγωνισμός λοιπόν στους καταναλωτές είτε σε επίπεδο νοικοκυριών είτε σε επίπεδο βιομηχανικό δεν είναι πολύ μεγάλη. Για την ολοκλήρωση της αγοράς η εικόνα είναι και εδώ ανακατεμένη λίγο. Θα δει κανείς ότι στη Βόρεια Ευρώπη έχει υπάρξει μια σύζευξη των συστημάτων των αγορών, όπως λέμε τεχνικά. Δηλαδή, ρυθμίζονται η προσφορά και η ζήτηση επί τη βάση ενός συστήματος λειτουργικού στα πλαίσια πολλαπλών χρηστών δικτύων. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μία μορφή ολοκλήρωσης της αγοράς η οποία δεν βασίστηκε μόνο σε θεσμικούς διακανονισμούς αλλά και στις επιθυμίες της ίδιας της βιομηχανίας. Απ' την άλλη όμως σε επίπεδο διαμεθοδιακής συνεργασίας υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αν κάποιος σαν παράδειγμα θέλει να αγοράσει φυσικό αέριο εκτός Πολωνίας και να το μεταφέρει στη Γαλλία, πρέπει να μισθώσει χωρητικότητα στους αγωγούς αναχώρα επί τη βάση διαφορετικών κανόνων, διαφορετικού κόστους σε κάποιες χώρες μέσω πληστηριασμών, χώρου σε άλλες χώρες μέσω άμεσων συμφωνιών, σε άλλες χώρες θα πρέπει να πληρώσει κανείς εκ των προτέρων την χωρητικότητα την οποία θα χρησιμοποιήσει, σε άλλες εκ των υστέρων, σε κάποιες χώρες πρέπει να το κοινοποιεί 5 το απόγευμα, σε άλλες 8 το πρωί. Συνεπώς λοιπόν υπάρχουν σημαντικές διαφορές και αυτό αυξάνει πάρα πολύ το κόστος της εμπορίας ενέργειας και εδώ μειώνονται νομίζω πολύ τα κέρδη και των παροχέων υπηρεσιών και του κοινού. Τι μπορούμε να κάνουμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν για να ολοκληρώσουμε την αγορά μέχρι το 2014. Πρώτον να εφαρμόσουμε πλήρως το λεγόμενο τρίτο πακέτο. Ενθυμίστε τις μακρότατες διαπραγματεύσεις η προθεσμία για την εφαρμογή της οδηγίας έληξε τον Μάρτιο του 2011 και μέχρι τον Ιούνιο δεν είχαμε δει και πάρα πολλές εφαρμογές από πλευρά των κρατών μελών. Τώρα τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Σήμερα το πρωί έλεγξα ότι οκτώ χώρες μας έχουν κοινοποιήσει πλήρη μεταφορή της οδηγίας, μεταφορά συγγνώμη της οδηγίας σε άλλες χώρες έχει ολοκληρωθεί σχεδόν η προσπάθεια αλλά δεν έχει κλείσει η διαδικασία και δεν έχουμε την τελική κοινοποίηση. Τέλος και σε επίπεδο ποιότητας βλέπω ότι έχουμε επενδύσει αρκετά σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε παράσχει τεχνική βοήθεια για αυτό το περίπλοκο νομοθετικό πακέτο. Νομίζουμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κακοφορία και η Ελλάδα και η Πορτογαλία είναι δύο από τις χώρες οι οποίες κοινοποίησαν πλήρη, πλήρη εφαρμογή του συστήματος και γενικά και οι χώρες αυτές βοηθούνται στα πλαίσια των ειδικών πακέτων και αυτή η προσπάθεια φαίνεται έχει κακοφορήσει. Εν πάση περιπτώσει παραμένουν δυσκολίες, υπάρχουν δύσκολες συζητήσεις στα κράτη-μέλη για διάφορα θέματα πολύ σημαντικά για την δημιουργία μιας συμπαγούς και ολοκληρωμένης αγοράς, όπως σαν παράδειγμα η ανεξαρτησία και οι αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών, όπως η απελευθέρωση ή καλύτερα αποδεσμοποίηση των αγορών. Λοιπόν, να πάω κάπως πιο γρήγορα τώρα. Να πω ότι πέραν της συνεχής παροχής τεχνικής βοήθειας προς τα κράτη-μέλη προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρως και τις δυνατότητες παρέμβασης επί παραλήψη τις οποίες έχουμε για μη κοινοποίηση, σαν παράδειγμα εφαρμογής μέτρων, για τη μη εφαρμογή μέτρων κτλ. Ένα δεύτερο σημαντικό συστατικό λοιπόν της εφαρμογής του τρίτου πακέτου είναι το θέμα της αποδεσμοποίησης, το θέμα του unbundling που έχει σαν στόχο να ξεχωρίσει την, προς, τα συμφέροντα αυτών που ασχολούνται με την προσφορά, με την διανομή. Από το 2007 και μετά ε, αυτή η κάθετη θα έλεγα ολοκλήρωση ήταν εμπόδιο για την εσωτερική αγορά και το τρίτο πακέτο λύνει το θέμα δημιουργώντας το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία του unbundling. Ε, βέβαια χρειάζεται μια διαδικασία η οποία προβλέπεται στο τρίτο πακέτο. Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να εγκρίνουν αναμία τις ε, προγραμματικές δηλώσεις των εταιριών που ασχολούνται με τη μεταφορά και θα έχουν την δυνατότητα επίσης να σχολιάσουν τις τελικές αποφάσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Ελπίζουμε να έχουμε τα τελικά στοιχεία τις επόμενες εβδομάδες, θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά έτσι ώστε να γίνονται σεβαστές οι προτάσεις μας. Αυτό που είναι δύσκολο στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας επικύρωσης είναι ότι μια θετική τάση γιατί κάποιες από τις κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις οι οποίες ήταν θα έλεγα κατά του unbundling για πάρα πολλά χρόνια έχουν αρχίσει να αλλάζουν θέσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Στη Γερμανία, σαν παράδειγμα, ανακοινώθηκε από μια τέτοια εταιρεία κάποιες εθελοντικές ιδέες μεταφοράς και από ε, ε, δυνατοτήτων μεταφοράς ενέργειας. Αυτό θα βοηθήσει να αναδιαρθρωθούν οι η γενικού ή καθολικού συμφέροντος υπηρεσίες όπως η διανομή. Ακούγονται πολλά επιχειρήματα ότι σαν παράδειγμα η αποθεσμοποίηση προκαλεί ιδιαίτερα υψηλό κόστος και πολλοί επιχειρηματολογούν λέγοντας ότι τελικά δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα. Νομίζω ότι εμείς συνολικά θα πρέπει να προσπαθήσουμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σαν πολιτική να συνεχίσουμε εμείς να μιλάμε για τα πλεονεκτήματα τα οποία παρέχει η εφαρμογή των συστημάτων που προβλέπουν την αποδεσμοποίηση. Το τρίτο πακέτο αυτό εσωτερικής αγοράς είναι κάποια θεσμικά στοιχεία, η δημιουργία της ΕΣΑ όπως επίσης και της Ένωσης των παροχέων και αυτών που ασχολούνται με τη διαχείριση των δικτύων. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν σημασία και η ΕΣΑ τώρα έχει πλήρες προσωπικό. Οι υπεύθυνοι διαχειριστές των δικτύων ήδη συνεργάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό είναι θετικό. Πέραν της εφαρμογής του τρίτου πακέτου υπάρχει κι άλλο ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό για μας σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το οποίο ονομάζουμε εμείς ο σχεδιασμός της αγοράς επί τη βάση των κανόνων στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως. Ενθυμίστε ότι το τρίτο πακέτο δημιούργησε ένα νέο μέσο ε, οι κατευθυντήριες γραμμές δικτύου όπως λέμε, όπου μέσα περίπλοκων μηχανισμών συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΣΑ, στους διαχειριστές του δικτύου και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί τη βάση ε, ιδίων κωδικών θα έλεγα. Η ΕΣΑ έχει ήδη οδηγήσει σε τρεις από τις πρώτες αυτές κατευθυντήριες γραμμές η Άνσος, δηλαδή ε, ε, οι συνδυασμένοι διαχειριστές δικτύου ε, προσπαθούν και αυτοί να προχωρήσουν. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει και ελπίζω ότι το 2014 θα έχουν ολοκληρωθεί οι προσπάθειες. Υπάρχουν παρόλα αυτά δυσκολίες και προκλήσεις. Κάποιες παλιές χώρες, όλες οι χώρες μάλλον, θα πρέπει να εγκρίνουν τις αποφάσεις αυτές σε επίπεδο επιτροπολογίας πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα ενιαίο ευρωπαϊκό γιατί αυτό θα μειώσει το κόστος και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Παρόλα αυτά όμως πιστεύουν ότι το δικό του σύστημα είναι αυτό που θα πρέπει να υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε συζητήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στην τελική φάση της προσπάθειας ε, για τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της αγοράς στο τομέα της ενέργειας και αυτή η απόφαση θα οδηγήσει σε επιπλέον νομοθετικές ρυθμίσεις δευτερευούσης σημασίας που θα πρέπει βέβαια όλες αυτές να ισχύσουν το ταχύτερο δυνατόν. Αυτά τα δύο σημεία λοιπόν. Πρώτον ότι το τρίτο πακέτο το οποίο έγινε καρπός τόσο δύσκολης διαπραγμάτευσης εφαρμόζεται πλέον και μπορούμε να περάσουμε στην πρακτική, ε, στην απελευθέρωση της αγοράς <coughs> και δεύτερον να δημιουργήσουμε κάποια ευρωπαϊκά πραγματικά συστήματα λειτουργίας των δικτύων και οργάνωσης των αγορών. Αυτοί είναι οι στόχοι τους οποίους έχουμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πετύχουμε τον δύσκολο αυτό στόχο για τις εσωτερικές αγορές. Αυτό φυσικά γίνεται και με το πακέτο για τις υποδομές. Έχει υπάρξει μια συζήτηση ξεχωριστή. Δέχομαι και ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, αν και δεν είναι τόσο δική μου αρμοδιότητα. Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας είναι κάτι το δύσκολο. Πάρα πολλά μένει να γίνουν, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες μπροστά μας, αλλά είναι κάτι το εφικτό, δεν είναι κάτι το μη ρεαλιστικό. Πολλά θα εξαρτηθούν από τη δυναμική της ε, ε, βιομηχανίας. Αν υπάρχει μια δυναμική η οποία διαπιστούνται σήμερα κάποιων επιχειρήσεων οι οποίες πραγματικά αποχωρούν ή μάλλον παίρνουν αποστάσεις από τον τομέα της παροχής και ασχολούνται με τη διαχείριση των δικτύων, τότε περνάμε στην ευρωπαϊκή αντίληψη για τη διαχείριση αυτών των ίδιων των δικτύων. Και όταν βλέπουμε κάποιες εταιρείες οι οποίες ήταν κάθετα ολοκληρωμένες θα έλεγα και οι οποίες μέχρι τώρα συστηματικά υπερασπιζόντουσαν το status quo και δεν έβλεπαν την, τον ανταγωνισμό σαν μια δυνατότητα, ενώ τώρα κάνουν κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή, αυτό δείχνει ότι μπορεί να κινηθούμε προς μια ανταγωνιστική αγορά. Πολλά θα εξαρτηθούν επίσης και από τις εθνικές πολιτικές στον τομέα της ενέργειας θέματα διασφάλισης ε, θα έλεγα ε, προμήθειας ενέργειας. Αν αντιμετωπίζονται αυστηρός εθνικά ε, θα δημιουργηθούν προβλήματα. Σαν παράδειγμα θα υπάρξουν προσπάθειες από κάθε χώρα αποθήκευσης ενέργειας σε αυστηρά εθνικό επίπεδο ή θα υπάρξει συνδυασμός της προσπάθειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι αποφάσεις για το λεγόμενο energy mix και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για να επηρεαστεί το λεγόμενο energy mix που είναι αρμοδιότητα φυσικά των κρατών μελών. Θα το κάνει κάθε χώρα μεμονωμένα ή θα λάβει υπόψη τις επιπτώσεις τέτοιων μέτρων στην λειτουργία της αγοράς και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Για όλα αυτά λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε τις ανταλλαγές εμπειριών ανάμεσα στις διάφορες χώρες Οργανώσαμε μια συνάντηση στις 20 Ιουλίου ανάμεσα στους Γενικούς Διευθυντές των Αρμόδιων Αρχών για να δούμε τι θα συνέχεια θα δοθεί ε, στις, ε, στην κατάσταση που δημιουργήθηκε στη Φουκουσίμα κτλ. Είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί και από τους Υπουργούς Ενέργειας ε, στο τέλος Σεπτεμβρίου και θα υπάρξει και μια διάσκεψη για την αγορά ενέργειας στις 29 Σεπτεμβρίου για τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος. Η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σαν στόχο τη διευκόλυνση των συζητήσεων και των ανταλλαγών απόψεων έτσι ώστε να εκτιμηθούν και οι συνέπειες των μέτρων αυτών σε κάθε χώρα και να έχουμε στη διάθεσή μας ε, κάποιες απόψεις για τα μέτρα τα οποία θα επηρεάσουν το λεγόμενο energy mix και πώς ε, τα μέτρα αυτά θα δημιουργήσουν ε, θετικές συνθήκες για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Αυτή ήταν η εισαγωγική παρουσίαση που έκανα από την πλευρά μου. Θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις, σκέψεις και ίσους ερωτήσεις. Κυρία Πέρνα, σας ευχαριστώ θερμά. Ε, ο συνάδελφος Φόποτα έχει, θέσει την πρώτη, έχει ζητήσει το λόγο για να κάνει την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Ε, δεν έχω καταλάβει αν είναι μισό άδειο ή μισό γεμάτο το ποτήρι. Πάντως ε, σίγουρα δεν είναι αρκετά γεμάτο. Ε, έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Εγώ είχα αρκετέ επικρίσεις όσον αφορά κάποια ακραία αιτήματα όσον αφορά την αποδέσμευση. Υπάρχουν κάποιες ενεργειακές εταιρείε, οι οποίες είναι πολύ περήφανε που έχουν ήδη εφαρμόσει την αποδέσμευση ή που ε, το κάνουν ε, αυτή τη στιγμή. Ε, Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουν την υποστήριξη του Κοινοβουλίου ε, και μάλιστα κατά των χωρών ε, που δεν έχουν εφαρμόσει επαρκώς το μέτρο αυτό. Ε, όσον αφορά τους ρυθμιστές, κάποιες χώρες δεν έχουν ρυθμιστές με αρκετή αρμοδιότητες. Και νομίζω ότι είναι σαφής η κατάσταση. Να επενδύσει κανείς σε γειτονική χώρα σημαίνει ότι πρέπει να ξεπεράσει σημαντικά εμπόδια. Και εάν υπάρχουν πολιτικοί και πόσο μάλλον κομματικοί παράγοντες, ε, αυτό νομίζω μπορεί να αποτρέψει αρκετούς από τις επενδύσεις. Θα πρέπει λοιπόν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να είναι ανεξάρτητες. Όσον αφορά την υποδομή, θα ήθελα να πω και εδώ κάποια λόγια, γιατί ιδιαίτερε εποχές όπως τις δικές μας, όπου χρειαζόμαστε επιγόντως ευρωπαϊκά επενδυτικά έργα, όπου θέλουμε επενδύσεις για την Ευρώπη με την ε, πραγματική σημασία της ε, λέξης, ε, θα πρέπει να πετύχουμε αύξηση των επενδύσεων. Και όσον αφορά τις αποφάσεις μεμονωμένων χωρών, όσον αφορά την πυρηνική ή όχι ενέργεια κλπ. άσχετα από αυτές χρειαζόμαστε επιγόντως επενδύσεις στην ενέργεια. Εάν ε, θέλουμε να μεταφέρουμε την ενέργεια και στο κέντρο της Ευρώπης, ε, χρειαζόμαστε την απαραίτητη υποδομή. Η υποδομή, λοιπόν, ε, είναι ένα μέσο ολοκλήρωσης της Ευρώπης, δημιουργίας της εσωτερικής αγοράς και όσον αφορά την αποθήκευση της ενέργειας, τη δέσμευση της ενέργειας, και αυτή μπορεί να επιτρέψει την ύπαρξη μιας πραγματικής διασυνοριακής συνεργασίας. Όσον αφορά τις προτάσεις για την υποδομή, υποβάλλατε κάποιες προτάσεις και άλλες προτάσεις εκπονούνται. Σημαντικό είναι ήδη από την αρχή η υποδομή αυτή να είναι ευρωπαϊκή. Και ε, να γίνει σωστή σύνδεση ανάμεσα στις διάφορες ε, μορφές ενέργειας. Συμπέρασμα λοιπόν, υποστήριξη για τις προσπάθειες ε, της Κομισιόν ε, να κινητοποιήσει τα κράτη-μέλη να κάνουν τα απαραίτητα βήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών. Και δεύτερον, όσον αφορά τις επενδύσεις, ως ε, μέσο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ε, θα πρέπει να προωθηθούν. Ε, ευχαριστώ ο συνάδελφος Κλάντε. Ναι, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Σπόμποτα. Οι εξελίξεις είναι τέτοιες που είναι σίγουρα αξιέπαινη η προσπάθειά σας. Προσπαθώ να τα πιστέψω όμως όλα αυτά. Μετά την Φουκουσίμα είδαμε ε, τις κυβερνήσεις ξαφνικά να θέλουν να εγκαταλείψουν την πυρηνική ενέργεια. Ε, στο μεταξύ όμως ε, αυτή αντιπροσωπεύει το 20% της συνολικής ενέργειας. Θα πρέπει να έχουμε την υποδομή για ε, αποθήκευση της ενέργειας. Ε, ε, στη Βάδη Βιρτεμβέργη η Βάτενφαλ εξετάζει τη δυνατότητα δέσμευσης. Δεν γίνεται ακόμα, εξετάζεται το θέμα αυτό. Κάθε ομοσπονδιακό κρατήδιο στη Γερμανία μπορεί μόνο του να αποφασίσει αν θέλει να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα αποθήκευσης της ενέργειας ή όχι. Μέχρι να ληφθεί η απόφαση μπορεί να μην μας ενδιαφέρει πια το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση. Και όταν ακούω ότι θέλετε έργα ε, που να ενισχύουν την εσωτερική αγορά ενέργειας, ε, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν διάφορα σχέδια για την ε, μεταφορά της ενέργειας στο τελικό καταναλωτή. μια μεγάλη επιχείρηση μπορεί να συναντά δυσκολίες ε, λόγω των ε, μεγάλων εκπομπών. Θα πρέπει να εξετάσει κανείς αν ε, θα πρέπει να λαμβάνουν άδειες για πραγματοποίηση των σχεδίων τους ή όχι. Είναι εύκολο να πούμε ότι το ενεργειακό μίξ, ο συνδυασμός των διαφόρων μορφών ενέργειας είναι θέμα του κάθε κράτους μέλους. Ε, θα πρέπει όμως ε, να δούμε αν θα καταλήξουμε τελικά σε ένα ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα. Κάποιοι μιλάνε για οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Ευρώπη, ε, άλλοι πηγαίνουν προ άλλη κατεύθυνση. Νομίζω πάντω ότι υπάρχουν πολλέ δυνατότητε για το μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ενημέρωση για όλα αυτά τα θέματα. Μιλήσατε για το διαχωρισμό μεταξύ προμήθειας και μεταφοράς. δεν μιλήσατε αρκετά για τις υποδομές και καταλαβαίνετε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα αυτά. Αυτό ενδιαφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μετά το διαχωρισμό που επιβλήθηκε αυτό το unbundling και από τότε που οι ιστορικοί άλλαξαν τους ισολογισμούς τους. Δεν μπορούμε να εντοπίσουμε πια τον ιδιοκτήτη των υποδομών, τον υπεύθυνο. Λέμε ότι η ρυθμιστική αρχή καθορίζει τις τιμές, αλλά ποιος αποφασίζει για τις επενδύσεις. Μήπως λοιπόν έγινε και η ώρα ώστε με πολύ μεροτρόπο τρόπο ο ιδιοκτήτης των υποδομών να κάνει μια αποτίμηση του συνόλου των υποδομών, μια ενημέρωση των υποδομών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, γιατί αυτή τη στιγμή εμπίπτει στον ιδιωτικό τομέα που είναι ρυθμισμένο. Τι θα γίνει αν η Gazprom έρθει και αγοράσει ένα σημαντικό τμήμα των υποδομών φυσικού αερίου. Λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει επιτήρηση από τις ρυθμιστικές αρχές. Θα δημιουργηθεί όμως πρόβλημα. Ε, τουλάχιστον ε, ε, θα είναι αρνητική εντύπωση στους πολίτες. Ποια είναι η γνώμη σας για τις υποδομές και ποιο είναι το μακροπρόθεσμο όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την πρόταση να διαβεβαιώσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες όπου, όπου και βρεθούν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια θα έχουν καλή, καλές υπηρεσίες και ποσοτικά και ποιοτικά σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Επίσης μιλήστε για ένα κεντρικό σταθμό αγοράς φυσικού αερίου στη, από την περιοχή της Κασπίας. Υπάρχει τέτοια πρόταση Υπήρχε πρόταση και παλιότερα που δεν βοδόθηκε όμως. Τι γίνεται, ποια είναι η, γνω... ποια είναι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το να δημιουργηθεί μια, ένα γραφείο αγοράς ε, φυσικού αερίου στην περιοχή της Κασπίας θάλασσας. Κυρία Μαδουρέλ, ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εξηγήσεις που μας έδωσε και συνεχίζοντας ε, τις παρατηρήσεις των συναδέλφων, θα ήθελα και εγώ να επιμείνω στην πιο διεξοδική ανάλυση του θέματος των υποδομών, που είναι απαραίτητο στοιχείο της ολοκλήρωσης της αγοράς. Γιατί είναι αδύνατο να ε, υλοποιήσουμε η ολοκλήρωση της αγοράς χωρίς να απαλείψουμε αυτούς τους, ε, αυτές τις ενεργειακές νησίδες. Γιατί δημιουργούν ε, πραγματικά στενοπούς και αυτή την απομόνωση ορισμένων περιοχών θα πρέπει να την εξαφανίσουμε. Μόνο έτσι θα υλοποιήσουμε μια πραγματικά ολοκληρωμένη ενεργειακή αγορά. Μην ξεχνάτε ότι ακόμη ένα τρίτο των χωρών μελών δεν έχουν υλοποιήσει το στόχο του 10% ε, δυναμικού διασύνδεσης, που ήταν ο στόχος που θέσαμε το 1992. Από αυτή την άποψη θα πρέπει επιτέλους να αναλάβουμε τη δέσμευση. Αυτός ο στόχος του 10% να θεωρηθεί το ίδιο, ο το ίδιο σημαντικός, το ίδιο σημαντικός με τους στόχους, ε, με το στόχο για τα 3-20%. Τις τρεις φορές ε, το 20% να θεωρηθεί εξίσου σημαντικός και ο στόχος του 10%. Ε, νομίζω ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την απόλυτη διακριτική ευχέρεια στα κράτη-μέλη για την, για, για την ενεργειακή ασφάλεια. Ούτε θα πρέπει να στηρίζεται αυτή μόνο σε αμυγός ε, εμπορικά κριτήρια. Βέβαια έγιναν κάποιες πρόοδοι στο θέμα αυτό, αλλά διαπιστώνουμε ότι μετά την πρώτη αποτίμηση του προηγουμένου Ιουνίου διαπιστώσαμε ότι λείπει αυτό το ευρωπαϊκό όραμα. Ερωτώ λοιπόν, δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να συμπληρώσουμε αυτή την εστίαση με μια πιο συγκροτημένη προσέγγιση που θα δίνει περισσότερη έφαση στην ευρωπαϊκή προοπτική. Ευχαριστώ. Κύριε Τζαβέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την κυρία Περνάετ για την παρουσίαση της εδώ. Ε, θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στην πιθανότητα δημιουργίας ενός hub center που θα φέρνει το αέριο από την Κεντρική Ασία. Σε αυτή την περίπτωση γνωρίζουμε ότι η Μπότας, η τουρκική εταιρεία ενέργειας, δεν δέχεται ε, για τη διέλευση, αλλά αλλάζει, βάζει το λεγόμενο καπέλο στην αγορά, ε, αλλάζει την τιμή του εισαγόμενου προϊόντος. Αν αυτό γίνει όπως καταλαβαίνετε δεν βοηθάει σε τίποτα να έχουμε το Hub Center γιατί θα πρέπει να πληρώνουμε αυξημένα διόδια σε εισαγωγικά στην Πότας. Χώρα διέλευση η Τουρκία, η Πότας είναι η, η τουρκική εταιρεία ηλεκτρισμού η οποία βάζει συνεχώς αυτά τα καπέλα για όποιον θέλει να εισάγει αέριο από την Κεντρική Ασία ή από το Ιράκ ή από το Τουρκμενιστάν. Αυτή είναι μία μου ερώτηση. Και η δεύτερη αφορά το security. Αναφερθήκατε ότι ε, τα κράτη-μέλη μεριμνούν για να υπάρξουν και κάποια ασφάλεια στην προμήθειά τους σε ενέργεια κτλ. Από άλλες πηγές είπατε. Ποιες άλλες πηγές εννοείται το shale gas, εννοείται κοιτάσματα αερίου που έχουν βρεθεί στο βόρειο μέρος της Ευρώπης και στο νότιο μέρος της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ε, Ο Πάουλ Ρούμπιχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις ε, διακόπες ήμουνα στην Κύπρο και εξέτασα εκεί την ε, ενεργειακή κατάσταση. Το θέμα της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ε, είναι ένα θέμα που τίθεται και εάν είναι δυνατή η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων δικτύων. Για τα νησιωτικά κράτη. Ε, η Κύπρος ε, είχε σημαντικά προβλήματα στην ενέργεια και η αγορά λόγω καταστροφής μέρους της υποδομής της. Ε, για παράδειγμα, στις ώρες αιχμής θα πρέπει όλοι, όλες οι βοηθητικές γεννήτριες ε, να βρίσκονται σε λειτουργία. Ε, αυτή τη στιγμή από την Αμερική και από πολλά άλλα μέρη υπάρχει ενδιαφέρον για την αγορά ενέργειας στην Κύπρο. Ε, η Κύπρος αυτή τη στιγμή από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχει τις περισσότερες ε, ώρες ηλιοφάνειας. Ε, στην Κύπρο, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν έργα ηλιακής ενέργειας. διότι υπάρχει τόση ηλιοφάνεια και μάλιστα ε, ε, είναι πολύ ε, οικονομικές οι τιμές των φωτοβολταϊκών κυψελών αυτή τη στιγμή σε όλη τον κόσμο. Μήπως θα είχε νόημα μια σχετική πρωτοβουλία της Κομισιόν στο, στην περιοχή αυτή. Η συνάδελφος Ρωμάνα Σιζίκ. Σας ευχαριστώ. Συζητήσαμε το πώς θα εντάξουμε τις εθνικές ενεργειακές πολιτικές στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Αυτό το ζήτημα δεν είναι μόνο πολιτικό, αλλά και τεχνικό, γιατί θα πρέπει να εκπληρωθούν πολλές τεχνικές προδιαγραφές και διάφοροι νόμοι της φυσικής. Το θέμα δεν είναι μόνο πολιτικό και τεχνικό, αλλά είναι και κοινωνικό-οικονομικό. Και οι επιλογές των μεμονωμένων χωρών είναι σημαντικές για το εθνικό επίπεδο. Αν ένα κράτο αποφασίσει να εφαρμόσει ρηξικέλευθε αλλαγέ στην ενεργειακή πολιτική του, ε, μια τέτοια απόφαση θα έχει αντίκτυπο και στην ενεργειακή αγορά γενικώ και στι γειτονικέ χώρε σίγουρα. Για παράδειγμα, έχω στο μυαλό μου τη Γερμανία αλλά υπάρχει και ένα γενικό ζήτημα που επισημαίνουμε εδώ. Στις συζητήσεις αυτές χρειαζόμαστε και μία αξιολόγηση για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν τις αποφάσεις τους σε ορισμένες χώρες και πού φτάνουν τα όρια της επικουρικότητας και της εθνικής κυριαρχίας για τέτοιου είδους αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής. Γιατί διαπιστώνουμε ότι στην Ευρώπη έχουμε τεράστια προβλήματα, ακριβώς επειδή είναι δύσκολο να ε, έχουμε τόσα εργοστάσια και το πού θα εγκατασταθούν. Θα πρέπει να βρούμε κατάλληλους χώρους για την ε, κατασκευή τέτοιων εργοστασίων. Ε, δεν θα πρέπει να μελούμε και τον προβληματισμό των πολιτών. Έλλειμμα υποδομών μεταφράζεται και σε έλλειμμα, έλλειψη ενεργειακών προϊόντων. Και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στους πολίτες. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έχω την ακόλουθη ερώτηση. Πού πιστεύετε ότι βρίσκονται τα όρια της κυριαρχίας των διαφορών χωρών και ποια θα πρέπει να είναι η συμβολή των χωρών για την σταθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς. Όλα αυτά τα στοιχεία ελήφθησαν δεόντως υπόψη θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση. Κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να στήσω συγγνώμη που έφτασα λίγο αργά και δεν ε, άκουσα όλη σας, ε, όλη σας την παρέμβαση. Ε, εάν ε, λοιπόν πρόκειται για πράγματα που ήδη έχετε πει θα μπορούσα να τα συζητήσουμε διμερώς, διότι δεν, ήθελα, δεν θα ήθελα να κουράσω τους συναδέρφους. Ε, Έχουμε πει ότι μας ενδιαφέρει η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Ε, τώρα, όταν κοιτώ την κατάσταση εντός των κρατών μελών, βλέπω ότι απέχουμε μίλια από τον στόχο μας. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη όπου υπάρχουν εθνικά μονοπόλια, υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν έχουν κάνει τίποτα Μπορεί νομοθετικά να γίνονται κάποια πράγματα, αλλά πολιτικά όσον αφορά το καθεστώς διοκτησίας δεν γίνεται τίποτα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν μια ειλικρινή συζήτηση για το θέμα αυτό και όσον αφορά την αποδεσμοποίηση την οποία επένδυσε πολύ ως ε, το μέσο με το οποίο θα ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας της ε, Ευρώπης. Ε, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ειδικά αυτό το μέσο δεν είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Κλωτ Τούρμες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ελπίζω οι διακοπές να ήταν ωραίες ή τουλάχιστον να ξεκουραστήκατε. Θα είμαι λιγότερο σκεπτικιστής σε σχέση με αυτά τα οποία πετύχαμε τα τελευταία χρόνια. Εγώ είμαι εδώ από το 99 και είναι αλήθεια ότι το δεύτερο και το τρίτο πακέτο για την εσωτερική αγορά προκάλεσαν αυτό που θα έλεγα μια πολιτιστική αλλαγή. Όχι μόνο ενέργεια, όχι μόνο ηλεκτρισμός, αλλά η ενέργεια ήταν ουσιαστικά εθνικά μονοπόλια στο παρελθόν. Και γι' αυτό υπήρξε έτσι η δυνατότητα να εξευρωπαϊστεί, θα έλεγα, όλη αυτή η αγορά και στον τομέα του φυσικού αερίου Βέβαια σε πολλές χώρες είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουν, ε, είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουν γρήγορα. Αλλά υπάρχουν θετικά και ένα από τα θετικά, τουλάχιστον για μένα, μια ότι μου είπαν ορισμένοι Γερμανοί φίλοι, συνάδελφοι και εμπειρογνώμονε ότι το λεγόμενο, η λεγόμενη αποχώρηση πυρηνική των Γερμανών θα ήταν δύσκολο να υποστηριχθεί πολιτικά αν δεν υπήρχε αυτή η αποδεσμοποίηση. Γιατί αν δεν υπήρχε η αποδεσμοποίηση, αυτοί οι οποίοι ήταν διαχειριστές των πυρηνικών εγκαταστάσεων θα είχαν και την ιδιοκτησία της πληροφόρησης για την κατάσταση του δικτύου. Το ότι υπήρξε η αποδεσμοποίηση και ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, αυτό οδήγησε στο αποτέλεσμα και για τη ρυθμιστική αρχή και για τους ε, λειτουργούς του δικτύου να μπορούν να πούν ότι έχουμε εντάσεις, έχουμε διαφορές, αλλά τις διαχειριζόμεθα. Πολλοί πιστεύουν το ότι ακριβώς επειδή αποδεσμοποιήσαμε την κατάσταση αυτή, αυτή την αγορά, έδωσε την πολιτική δυνατότητα στην κυβέρνηση να κάνει αυτή την αλλαγή. Πετύχαμε λοιπόν μεγαλύτερη διαφάνεια πετύχαμε μεγαλύτερη ανεξαρτησία για τους εμπλεκομένους. Μια άλλη ιδέα την οποία προώθησε ο κύριος Σοντή είναι το πόσο αυτό το δίκτυο μπορεί να λειτουργήσει διεθνικά. Η ιδέα την οποία εκφράσατε για να υπάρξουν περισσότερα κοινά διεθνή και ευρωπαϊκά στοιχεία ολοκλήρωσης της αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Η ιδέα είναι καλή, ας μην είμαστε απεσιόδοξοι. Δείτε σήμερα το τι γίνεται ανάμεσα στην αγορά του Μπενελούξ και τη Γερμανία. Έχουμε μια εταιρεία η οποία λειτουργεί στην Ολλανδία, στη Βόρεια Θάλασσα και φτάνει και στην, στα σύνορα της Αυστρίας. Και υπάρχει σύνδεση της υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Αυστρία που παρέχει ηλεκτρισμό στη Γερμανία. Και για το φυσικό αέριο έχουμε επίσης εταιρείε δραστηρίες στην Ολλανδία, στη Γερμανία ταυτόχρονα κτλ. Έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε την εθνική διάσταση. Και όπως είπε ο κύριος Σοντή θα πρέπει να συνεχίσουμε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση έτσι ώστε να καταφέρουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Κάποιες ερωτήσεις προς την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτον, αν πράγματι θέλουμε περιφερειακή ολοκλήρωση σε σχέση με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τότε θα πρέπει οι ρυθμιστικές αρχές αναχώρα των χωρών να συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους. Εγώ δεν έχω πάρει απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γύρω από αυτό. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να διευκολύνει ότι η ρυθμιστική αρχή της Γερμανίας, της Ισπανίας, του Βελγίου κτλ. κτλ να ασχολούνται τα θέματα όχι μόνο στην Βόρεια ή στη Βορειοδυτική Ευρώπη αλλά εν πάση περιπτώσει μια κάποια πραγματικότητα της αγοράς να αντικατοπτρίζεται σε αυτή τη μορφή συνεργασίας. Εάν ο διαιτητής δεν είναι υπερεθνικός, πώς μπορούμε να περιμένουμε από τους παίκτες να είναι υπερεθνικοί. Λοιπόν, η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και πίεζε έτσι ώστε να υπάρξει περισσότερος ανταγωνισμός στη χονδρική αγορά. Είχε υπάρξει και η υπόθεση την οποία ανέλησε η Γενική Διευθύνση Ανταγωνισμού και έχω την εντύπωση, υποκειμενική βέβαια, ότι από τη σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη προθυμία έτσι ώστε να παρακολουθούν την εύρυθμη λειτουργία των αγορών και κατά πόσον λειτουργούν σωστά οι αγορές. Να μην ξεχνάμε ότι για την ανταγωνιστικότητα των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ο, ο, βασικός, ο, ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει τα πράγματα είναι η εύρυθμη λειτουργία σε εθνικό επίπεδο. Ξέρουμε ότι το κόστος φτάνει και τα 30 ευρώ το ΜΒ. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθήσει πολιτικά να βοηθήσει την κατάσταση. Σας ευχαριστώ κυρία Φιγερέδο. Το Ευχαριστώ. Έχω και εγώ δύο ερωτήσεις που με απασχολούν σε αυτή τη διαδικασία δημιουργίας ή διεύρυνσης της εσωτερικής αγοράς. Ο πρώτος προβληματισμός μου αφορά τις διαφορές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Διαφορές όχι μόνο ως προς την κατάσταση των φορέων των παρόχων, αλλά και διαφορές ως προς τις υποδομές. Επίσης υπάρχουν διαφορές και στην οικονομική κατάσταση των χωρών μελών. Ανακύπτει λοιπόν το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε μία ανάπτυξη των υποδομών σε χώρες που αντιμετωπίζουν δεινά οικονομικά και δημοσιονομικά αλλά και κοινωνικά προβλήματα. Και πώς θα βοηθήσουν αυτές τις χώρες, πώς θα τις στηρίξουμε προκειμένου να εξυγχρονίσουν τις υποδομές τους και πώς θα εξασφαλίσουμε μια καλή κατανομή της ενέργειας ηλεκτρικής, φυσικού αερίου ή οποιασδήποτε μορφής. Η πρώτη ερώτηση ήταν αυτή. Η δεύτερη που είναι συναφής με την πρώτη αφορά τις τιμές της ενέργειας. Ποιε είναι οι τιμές που θα καταβάλουν οι τελικοί καταναλωτές. Είτε είναι αυτοί μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε είναι τα νοικοκυριά γιατί η αύξηση των ενεργειακών τιμών, η αύξηση των φόρων, όλες αυτές οι αυξήσεις ε, σε συνδυασμό με τις μειώσεις των μισθών που παρατηρούμε πολλές φορές ή με την ε, αύξηση της ανεργίας και με την όξη της φτώχειας, όλα αυτά οδηγούν σε μια ενεργειακή ένδυα. Ποια μέτρα λοιπόν θα προτείνουμε για να λάβουμε υπόψη αυτή την κατάσταση. Ή μήπω. αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι μια όξυνση των διαφορών και μια ενίσχυση των ανισοτήτων και στις υποδομές και στην κατανομή της ενέργειας αλλά και στην πρόσβαση στην ενέργεια. Μήπως εκεί οδηγούμαστε τελικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα επανέλθω σε ένα, σε ένα θέμα που επανειλημμένως αναφέρθηκε και από τους προλαλήσαντες, το θέμα των υποδομών και της απαραίτητης χρηματοδότησης αυτών των υποδομών. Γιατί πραγματικά οι υποδομές χρηματοδοτούνται ουσιαστικά από τις αγορές. Πρόσφατα, σε μια έκθεση, την έκθεση Σούζα Βάγνερ, υποβάλλεται προτάσεις για τις ενεργειακές υποδομές και έχουμε τέτοιες προτάσεις και για καινοτόμα χρηματοπιστωτικά εργαλεία ή κοινωνικά, κοινοτικά συγγνώμη, ενωσιακά ταμεία ή ε, προσφυγή στα κεφάλαια κινδύνου. Είχαμε υποβάλει μια σειρά τέτοιων προτάσεων συγκεκριμένων. Ποια είναι η θέση σας για τις προτάσεις αυτές της έκθεσης. Έχουμε και κάποια σχέδια υποδομών που μπορεί να έχουν θεμελιώδη σημασία, αλλά να μην είναι αποδοτικά ή κερδοφόρα. Θα τα αφήσουμε στη μοίρα τους, στο έλεος του Θεού. Θέλουμε μια συνεργασία βιομηχανίας και δημοσίων αρχών, ίσως με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού Πώς σκοπεύετε να ενθαρρύνετε τέτοιου είδους συγχρηματοδοτήσεις για τη βελτίωση των υποδομών. Η κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τις εμπειρίες που μετέφερε ο κύριος Ρούμπιχ και εγώ ε, έζησα κάτι στην Πολωνία το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για τις υποδομές. Υπήρξε μια διακοπή στην παροχή ενέργειας κάθε φορά που έβρεχε. Νόμιζα ότι ήταν όπως ε, τότε με τον κομμουνισμό, όποτε έβρεχε τότε σταμάταγε και το, ο ηλεκτρισμός στο σπίτι. Διαρωτώ με λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα των υποδομών για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αν πράγματι χρειαζόμαστε μια ουσιαστική εσωτερική αγορά, απαιτεί το εξυγχρονισμό των δικτύων κάθε χώρας. Γιατί αν κάθε φορά που πέφτει ένα δέντρο ή ο άνεμος δημιουργεί προβλήματα, δεν θα πρέπει να είμαστε μάρτυρες μιας τέτοιας ε, διακοπής της παροχής ρεύματος. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε έτσι ώστε να επιβάλλετε τον εξυγχρονισμό των υπαρχόντων δικτύων. Και δεύτερον θα ήθελα να υποστηρίξω τον συνάδελφο που μίλησε για την ιδιοκτησία. Έχω την αίσθηση ότι όταν συζητάμε για τα θέματα της ασφάλειας παροχής ενέργειας δεν γνωρίζουμε τι γίνεται με την ιδιοκτησία πολλών επιχειρήσεων. Το θέμα αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα δεν μιλάμε μόνο για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σόντι, αλλά το θέμα είναι ποιος αγοράζει σαν παράδειγμα στην Πολωνία τα δικαιώματα για την εξόριξη φυσικού αερίου, για την, μάλλον για την αναζήτηση φυσικού αερίου σε συγκεκριμένες περιοχές. Πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για την ιδιοκτησία των επιχειρήσεων που επενδύουν στον τομέα της ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να θέσω δύο-τρεις ερωτήσεις. Η Κομισιόν πώς εκτιμάει το δυναμικό θα ταιριάξει στην εσωτερική αγορά. Και δεύτερον, όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, θέλουμε μεγαλύτερο μερίδιο στην ε, αγορά. Ε, το μερίδιο όμως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εξάγονται αυξάνεται, το οποίο σημαίνει ότι μειώνεται το μερίδιο εντός της αγοράς. Και Πώς το βλέπει αυτό η Κομισιόν. Ε, κυρία Μπέρνας, ακούσατε πάρα πολλές ερωτήσεις. Μήπως μπορείτε να προσπαθήσετε να απαντήσετε στο βαθμό που είναι δυνατόν. Είναι πολύ ευρύ το θέμα. Ε, προσπαθήστε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ όλους για τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις σας. Χαίρομαι που βλέπω το ενδιαφέρον σας και τον βαθμό ανάλυσης ε, στον οποίο ενδιαφέρεστε να συζητήσετε τα θέματα αυτά. Να ξεκινήσω από το θέμα της ε, υποδομής. Νομίζω ότι λανθασμένα δεν το συμπεριέλαβα αυτό στην παρουσίασή μου, διότι πίστευα ότι οι πληροφορίες που έχετε στο θέμα αυτό είναι πιο αναλυτικές από ό,τι ε, για τα άλλα θέματα. Σίγουρα όμως η ολοκλήρωση της υποδομής, ε, η συμπλήρωση των ε, κενών, ο εξυγχρονισμός του δικτύου διανομής καθώς και τα ΦΙΗ δίκτυα, τα smart grids αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της ενίας, της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Χωρίς την ολοκλήρωση των δικτύων δεν μπορεί να υπάρχει διασυνοριακό εμπόριο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Η ε, Κομισιόν έχει ε, εκπονήσει μια ξεχωριστή στρατηγική για την υποδομή, ε, εξετάζει νομοθετικές προτάσεις, τις οποίες προτίθεται να υποβάλει Οκτώβριο ή Νοέμβριο. Νομίζω ότι αυτό θα καλύψει τέσσερα θέματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι τα βασικά σημεία που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όσον αφορά το πακέτο της υποδομής. Το πρώτο σημείο είναι ο προγραμματισμός της υποδομής. Αρκετοί από εσά ανέφεραν ότι η ανάπτυξη δεκαετών ε, προγραμμάτων ε, είναι πολύ σημαντική διότι ε, ε, έτσι υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική στην ανάπτυξη της υποδομής. Συμφωνούμε πολύ με την Κομισιο... Συμφωνεί πολύ η Κομισιόν με το θέμα αυτό και θέλουμε αυτό να αντικατοπτρίζεται στην πρότασή μας ότι οι εξελίξεις θα πρέπει να βασίζονται σε προγράμματα που ξεκινούν από την βάση. Ε, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι βασικοί διάδρομοι που θα πρέπει να αναπτυχθούν ε, εντό της Ευρώπης. Ε, το άλλο θέμα το οποίο έχουν τονίσει όλοι οι ενδιαφερόμενοι είναι οι δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τις διαδικασίες προγραμματισμού. Και αυτό αναφέρθηκε εδώ στην συζήτηση από τοπικές κοινωνίες που επηρεάζονται από τις επενδύσεις στις, ε, υποδομές, ε, στις υποδομές έχουμε ακούσει ε, σχετικές διαμαρτυρίες. Είναι και αυτό λοιπόν ένα θέμα το οποίο θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τα θεμητά ε, συμφέροντα των ε, τοπικών ε, κοινοτήτων αλλά να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε και τις διαδικασίες κατά την ανάπτυξη των προγραμμάτων. Η επόμενη φάση είναι να υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο που να επιτρέπει την, την επένδυση στην... Ε, στις ενεργειακές υποδομές. Ε, από τη φύση το θέμα αυτό συχνά είναι μονοπόλιο, γι' αυτό είναι σημαντικό όταν οι επενδυτές λαμβάνουν σχετικές αποφάσεις ε, να ε, γνωρίζουν ε, ότι με το σύστημα αυτό θα έχουν ένα δίκαιο κέρδος με βάση τις επενδύσεις που θα έχουν κάνει. Και τέταρτον και εμείς στην Κομισιόν ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει η αγορά να ε, χρηματοδοτήσει τις ε, επενδύσεις και μόνο όταν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό οι αγορές τότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δημόσιοι πόροι. Ε, διασφαλίζονται στον μέγιστο βαθμό δυνατό ε, ότι θα μπορέσουν ε, να αποτελέσουν μοχλό για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Θα ήθελα όμως επίσης να τονίσω ότι η διασφάλιση της ανάπτυξης της υποδομής δεν έχει να κάνει μόνο με την ανάπτυξη πρόσθετων υποδομών, έχει να κάνει και με την χρήση με την πιο αποτελεσματική χρήση ε, της υπάρχουσας υποδομής. Βλέπουμε ότι υπάρχει συμφόρηση σε πολλά σημεία της υποδομής, ε, μακροπρόθεσμα κιόλας. Ε, εάν γίνει όμως... Εάν εξετάσει κανείς την από τεχνικής άποψης ε, του ε, τους συνδέσμους ε, βλέπουμε ότι δεν έχει εξαντληθεί όλο, όλο το δυναμικό τους και έτσι από τεχνικής πλευράς δεν υπάρχει συμφόρηση. Φυσικά δεν θα πρέπει να επενδύσουμε στην ε, κατασκευή νέου αγωγού δίπλα σε έναν υπάρχοντα εάν δεν έχει εξαντληθεί ε, το δυναμικό του υπάρχοντος ε, αγωγού. Το επόμενο θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ έχει να κάνει με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής στην εσωτερική αγορά και με την και με τις θέσει σχετικά με την αποδοσμοποίηση. Συμφωνώ με τον κύριο Τουρμέ, ότι τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δεν είναι αποκλειστικά αρνητικά. Είχαμε και κάποια θετικά αποτελέσματα με την ε, απελευθέρωση του ενεργειακού τομέα. Εάν κοιτάξετε για παράδειγμα πώς, η, ε, πώς έχει αντιδράσει η αγορά φυσικού αερίου στην ε, δυτική Ευρώπη στις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά, διότι ε, λόγω των τιμών ε, ήταν ε, χαμηλή η ζήτηση και υψηλή η προσφορά. Αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο στις τιμές χονδρικής. Δυστυχώς δεν είδαμε παρόμοια δυναμική στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά εάν οι αγορές αλλά είδαμε ότι οι αγορές αρχίζουν και λειτουργούν. Άλλο παράδειγμα είναι η απόφαση της ε, Γερμανίας ε, να ε, διακόψει την πυρηνική παραγωγή ενέργειας. Αυτό είχε σημαντικό αντίκτυπο στη διαμόρφωση των τιμών. Εάν κοιτάξετε όμως την παρουσίαση που μας υπέβαλε η Γερμανία στην συνάντηση της 20ης Ιουλίου ε, θα είδατε ότι η αντίδραση στις τιμές ήταν πολύ βραχυπρόθεσμη. Αμέσως μετά ε, είδαμε ο ομαλοποίηση, ε, εξομάλυνση των τιμών. Οι αγορές λοιπόν λειτουργούν. Επίσης αν κοιτάξετε τη ρευστότητα στις αγορές αυτή αυξάνεται. αυξάνεται ο όγκος ε, και του ηλεκτρικού ρεύματος ε, και του φυσικού αερίου ε, που αποτελεί αντικείμενο εμπορίου. Όπως ανέφερα λοιπόν στην παρουσίασή μου, μπορεί να μην βλέπουμε αρκετό ανταγωνισμό όσον αφορά την παραγωγή ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Πολύ συχνά οι προμηθευτές ε, αγοράζουν ενέργεια από έναν βασικό προμηθευτή ε, σε κάποια χώρα. Θα πρέπει λοιπόν μαζί με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές να παρακολουθήσουμε την κατάσταση. Επίσης η λειτουργία των αγορών λιανικής είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω όσον αφορά την αποδεσμοποίηση. Δεν είμαι τόσο απεσιόδοξη, διότι αν κοιτάξετε τα νούμερα, τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν ζητήσει διαχωρισμό του καθεστώτος ιδιοκτησίας. Ιδιαίτερα όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, βλέπουμε πιο ισχυρή τάση από ότι στο φυσικό αέριο. Ε, πολλοί έχουν ε, επιλέξει αυτού του τύπου την αποδεσμοποίηση και ακόμα και σε κράτη-μέλη όπου υπάρχει ε, δυνατότητα επιλογής. Οι οικονομικοί φορείς επιλέγουν όλο και περισσότερο τον ε, διαχωρισμό του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Ε, αυτό λοιπόν είναι, είναι μια τάση που θα συνεχιστεί στο μέλλον. Ε, πιστεύουμε στο, στην απελευθέρωση αυτή των ε, φορέων ε, των ε, συστημάτων διαβίβασης όσον αφορά Βλέπουμε ότι ενεργούν όλο και πιο ανεξάρτητα οι φορείς αυτοί και όχι ως τα μικρά αδέρφια των μεγάλων επιχειρήσεων ενέργειας. αναφέρθηκαν διάφορα παραδείγματα ε, τέτοιων ε, φορέων ε, των συστημάτων διαβίβασης. Η Χέλια είναι ένας από αυτούς τους φορείς. Όπως ανέφερα στην παρουσίασή μου, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά τις εξελίξεις, ώστε άλλοι που διστάζουν περισσότερο είτε σε επίπεδο κράτους μέλους είτε σε επίπεδο επιχείρησης, θα πρέπει να φροντίσουμε οι ε, φορείς αυτοί να ε, συμμετάσχουν περισσότερο στον ανταγωνισμό. και να αλλάξουν την ε, επιχειρηματική τους νοοτροπία. Όσον αφορά τη διαφοροποίηση των ε, ενεργειακών πηγών. Ε, πολλές αναφορές έγιναν ε, στην Κασπία θάλασσα και στον Αγωγό Ανέφερα πριν ότι δεν βλέπουμε την ίδια τάση στην Ανατολική Ευρώπη που βλέπουμε και στην Δυτική Ευρώπη όπου είδαμε ότι η παγκόσμια δυναμική προσφοράς και ζήτησης έχει επηρεάσει πολύ τις τιμές. Η Ανατολική Ευρώπη είναι πιο εκτεθειμένη σε έναν μοναδικό προμηθευτή και δεν έχει την ε, δυνατότητα διαφοροποίησης στον τομέα αυτών. Όσον αφορά ε, τη δυνατότητα αποθήκευσης ε, θα πρότεινα την δημιουργία κέντρων για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και Στόχος ε, είναι να υπάρχει διαφοροποίηση της ε, προμήθειας ε, και στα κράτη-μέλη μέσω ενός κέντρου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Τα σχετικά κράτη-μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τα θέματα αυτά σε περιφερειακό επίπεδο έγινε πρόταση εμείς ως Κομισιόν ε, να κινητοποιήσουμε τους εθνικούς ε, ρυθμιστικούς φορείς ε, να συνεργαστούν και σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό νομίζω ότι είναι σωστό. Σε κάποιο βαθμό η περιφερειακή συνεργασία λειτουργεί αρκετά καλά όταν δούμε την αγορά ηλεκτρισμού στην Βόρεια Ευρώπη και αλλού. Ε, ωστόσο, συμφωνώ ότι η, η ίδια αυτή η στενή συνεργασία δεν υπάρχει ε, σε άλλες περιφέρειες, ούτε ε, υπάρχει στον τομέα του φυσικού αερίου. Ως Κομισιόν έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία ε, τον Απρίλιο ή τον Μάιο νομίζω ήταν ε, να ζητήσουμε μέχρι τον Ιούλιο οι εθνικές δημιουργικές αρχές να μας πούνε πώς θεωρούν ότι οι διάφορες περιφέρειες θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Ε, και έχουμε στοιχεία και για τον τομέα του ηλεκτρισμού, όχι μόνο για τον τομέα του φυσικού αερίου. Ελπίζουμε λοιπόν ότι και οι περιφέρειες ε, θα εκμεταλλευτούν τι δυνατότητε να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση τη ενιαία αγορά. Σε ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθεια, αναφέρθηκε και το θέμα των διαφόρων κέντρων προκειμένου να διευκολύνουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Δεν ξέρω βέβαια. Προηγουμένως αναφερθήκαμε στο κατά πόσο οι κρατικές αρχές θα πρέπει να ενεργήσουν ως εταιρείε ή ως επενδυτές. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη και διαλλακτική να εξετάσει και τις προτάσεις της βιομηχανίας, αλλά δεν αισθανόμαστε την ανάγκη εμείς να οργανώσουμε μια τέτοια δομή. Και μια τέτοια πρόταση της βιομηχανίας θα αξιολογηθεί με βάση τους κανόνες ανταγωνισμού. Γιατί αν γίνεται συλλογική αγορά αερίου, για παράδειγμα, από ε, σημαντικούς ε, προμηθευτές ενέργειας στην Ευρώπη, τι θα γίνει σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό μεταξύ τους ε, στην περαιτέρω πώληση αυτού του αερίου στην αγορά. Η το γεγονό τη συλλογική αγοράς μπορεί να μην, να μην δημιουργεί πρόβλημα, αλλά από άποψη ανταγωνισμού θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει κατόπιν με την πώληση αυτού του αερίου που έχει αγοραστεί συλλογικά. Θα πρέπει η βιομηχανία εδώ να μα υποβάλει μια πρόταση την οποία θα αξιολογήσουμε. Το θέμα της διαφάνειας επίσης απασχολεί πολλούς. Επιθυμία για μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία των δικτύων μεταφοράς ή της ιδιοκτησίας μεριδίων σε εταιρείε παραγωγής ενέργειας. Θέλουμε φυσικά στην ενέργεια διαφάνεια και εγώ προηγουμένως είχα απασχοληθεί στον τομέα τηλεπικοινωνιών και με σώκαρε αρχικά η αδιαφάνεια που διαπίστωσα στον τομέα της ενέργειας. Ήταν δύσκολο να ενημερωθούμε για το περιεχόμενο μακροχρόνιων ε, συμβάσεων, για τη δομή ε, της ε, συμμετοχής σε εταιρείε, των μεριδίων σε, μετοχών σε εταιρείε. Νομίζω ότι ως προς τη διαφάνεια έχουμε σημειώσει αρκετά ενθαρρυντικά βήματα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, άσκησε επιρροή σε ό,τι αφορά το σύστημα καταχώρησης των φορέων. Επίσης, κανόνες για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαφάνειας. Γιατί το πρώτο κριτήριο, η πρώτη ερώτηση που θα θέσουμε στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές όταν εξετάζουμε τη διαδικασία επιστοποίησης είναι μια λεπτομεριακή αναφορά του ποιο είναι ο ιδιοκτήτης αυτών των μονάδων μεταφοράς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη διαφάνεια πιστεύω. Σε ό,τι αφορά τις αγορές, το δυναμικό των αγορών, capacity markets. Αυτό το θέμα μας ε, απασχολεί εδώ και καιρό και αν οι αγορές αυτές μπορούν να χρηματοδοτήσουν ε, τις ε, απαιτούμενες επενδύσεις για την ηλεκτροπαραγωγή για παράδειγμα θα πρέπει να είμαστε διαλεκτικοί και ανοιχτόμυαλοι. Βέβαια, ο διάβολος καραδοκεί στις λεπτομέρειες. Τι γίνεται σε περίπτωση ανάγκης παρέμβασης στην αγορά. Όταν υπάρχει παρέμβαση στην αγορά θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα καταπνίξουμε τα θετικά ε, σημάδια που θα μπορούσε να μας δώσει η αγορά για το πού είναι αποτελεσματικές οι επενδύσεις. Και από τη στιγμή που ληφθούν κάποια μέτρα θα πρέπει να είναι αναλογικά, σωστά στοχευμένα και να μην έχουν αρνητικές ε, παρενέργειες και να μην ε, απομονώσουν μεγάλο τμήμα της προμήθειας ενέργειας και τα εξοβελήσουν από την αγορά. Για παράδειγμα, μιλήσαμε με την, με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πυρηνική ενέργεια. Τώρα, ποια είναι η αξία των διαφόρων δειγμάτων ε, τιμών. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταλήξει σε απάντηση, αλλά αυτό το θέμα σίγουρα θα πρέπει να το εξετάσουμε στην ανάλυση που θα κάνουμε για να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να αλλάξουμε το σχεδιασμό της αγοράς αν υιοθετήσουμε ένα νέο μοντέλο όπου μεγάλο τμήμα της παραγωγής θα προσανατολίζεται ε, σε μέτρα παρέμβαση της αγοράς. Σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση, τον καθορισμό των τιμών και το θέμα της ε, ενεργειακής ένδυας, η την αρνητική επιρροή που υφίστανται τα νοικοκυριά από την απελευθέρωση είναι αρκετά δύσκολο ζήτημα. Ακούσαμε το θέμα των blackout των διακοπών στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην Πολωνία. Και σίγουρα ε, δεν γίνονται αρκετές επενδύσεις στις υποδομές και στη συντήρησή τους. Γιατί θα πρέπει τα δίκτυα να είναι μονίμως σε καλή κατάσταση και να εξασφαλίζουν την προμήθεια στους καταναλωτές. Βέβαια, το θέμα των επενδύσεων είναι, λέτε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το θέμα των τιμών και της δυνατότητας που έχουν οι καταναλωτές να καταβάλουν συγκεκριμένη τιμή. Πολλές φορές το εισόδημα των νοικοκυριών επωφελείται και επηρεάζεται αυτές τις ρυθμισμένες τιμές. Θα πρέπει όμως να δούμε ποιο είναι το επίπεδο αυτών των τιμών και επηρεάζεται το επίπεδο των τιμών από το πόσο κοντά βρίσκονται οι αγορές ε, χονδρικής. Πάντως, ως Επιτροπή θα πρέπει και αυτό το θέμα να το προσέξουμε και εκκρεμούν κάποιες διαδικασίες επί παραβάση κατά κρατών μελών. Στόχος μας βέβαια δεν είναι να πούμε στα κράτη-μέλη ότι οι ρυθμισόμενες αυτές τιμές θα πρέπει εξορισμού να απαγορεύονται. Απλώς φροντίσουμε ώστε αυτές οι τιμές να είναι, ρυθμισμένες να είναι σωστά στοχοθετημένες. Γιατί άλλο είναι οι καταναλωτές που χρήζουν ειδική προστασίας από συγκεκριμένες ρυθμισμένες τιμές ελληνικής και άλλο οι καταναλωτές που ίσως δεν χρειάζονται τέτοιου είδους προστασία. Γιατί όσο αναπτύσσονται η αγορά και ο ανταγωνισμός θα πρέπει του, τις ρυθμίσεις για τις τιμές να τις ε, επικεντρώνουμε μόνο στη, στα πιο, στους πιο ευπαθείς καταναλωτές που χρειάζονται τέτοιας ενίσχυσης. Και σε περίπτωση μόνο που αυτό, αυτό είναι το μόνο μέτρο που θα βοηθήσει τους καταναλωτές που πλήττονται από την ε, ενεργειακή ένδυα. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως άλλα μέτρα μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά από τις ρυθμισμένες τιμές. Κάποιες χώρες ε, προσέχουν υπερβολικά ε, σε αυτό το θέμα των αριθμισμένων τιμών για να υιοθετήσουν, ε, για να υλοποιήσουν αυτό το στόχο. Και νομίζω ότι η γενικευμένη χρήση των αριθμισμένων τιμών έχει αρνητικά αποτελέσματα, γιατί δημιουργεί αρνητικό κλίμα και για τις επενδύσεις. Δεν ξέρω αν παρέλειψα κάποιες ερωτήσεις. Φοβάμαι ότι δεν ε, κάλυψα όλα τα θέματα. Αν μου διέφυγε κάποια ερώτηση, παρακαλώ να μου την υπενθυμίσετε. Αλλά μπορούμε και διμερώς να επικοινωνήσουμε και να σας στείλω τις απαντήσεις. Να σας ευχαριστήσω θερμά κυρία Μπέρναρτς. Πολλές ερωτήσεις ακούσαμε, πολύ αναλυτικές απαντήσεις. Σας ευχαριστώ θερμά και νομίζω θα δεχτούμε την πρότασή σας. Θα ήταν χρήσιμο να λάβουμε έναν κατάλογο, όχι μια ογκώδη μελέτη, αλλά έναν κατάλογο των προβλημάτων ε, αναχώρα. Ε, θα σας στείλουμε και γραπτό αίτημα. Θα ήταν χρήσιμο αυτό για να αποκτήσουμε μια καλή εικόνα. Να σας ευχαριστήσω θέρμα ε, για την επισκεψή σας, για τη συζήτηση αυτή. Και έτσι κλείνουμε το θέμα υπαριθμών 5 στην ημερήσια διάταξη και περνάμε έτσι στο πρώην 4 νυν 6 της ημερήσιας διάταξης.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 it works. Well, somebody told me that it should. Oh, wonderful. Okay, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, περνάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο σημείο, το σημείο 6. Και θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Πριν. που αντιπροσωπεύει την ομάδα υψηλού επίπεδου για τις συγκεκριμένες αυτές ένα θέμα εν πάση περιπτώσει πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας, έχετε το λόγο. Και σας θυμίζω ότι έχουμε και μια δημοσίευση εδώ, πολύ ενδιαφέρουσα, την οποία μπορείτε να κοιτάξετε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους, διότι ωστέ Εξ ονόματος της ομάδας εμπειρογνωμόνων Υψουλού επίπεδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2010, έχετε όλη την έκθεσή μας, την παρουσιάσαμε τον προηγούμενο μήνα. θα ήθελα να αναφερθώ στα βασικά χαρακτηριστικά της έκθεσης αυτής και να ζητήσω τη στήριξή σας για την εφαρμογή των προτάσεων. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να προκαλέσει ενδιαφέρον Θα δείτε άλλωστε ότι οι εμπειρογνώμονες οι οποίες πήραν μέρος στη σύνταξη της έκθεσης αυτής είναι σημαντικές προσωπικότητες των νέων τεχνολογιών, όλων των τομέων και λέγουν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα σύντομα σε κάποιους τομείς γιατί τότε αν δεν ληφθούν μάλλον τότε δυστυχώς πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης κινδυνεύουν να χαθούν στις εκλογικές σας περιφέρειες ιδιαίτερα σε προχωρημένες τεχνολογίες της κατασκευαστικής βιομηχανίας, της έρευνας και της ανάπτυξης. Γενικά πάρα πολλές θέσεις εργασίας θα απολεστούν σύντομα. Θα πω λίγα λόγια εισαγωγικά και θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας αν επιθυμείτε. Θα ήθελα να αναφερθώ να κάνω ένα απολογισμό του τι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και να πω επίσης και ποιες είναι οι προτάσεις οι οποίες γίνονται. Τομείς όπως η βιοτεχνολογία, η μικροεκλεκτρονική, η φωτονική, όπως επίσης και η μικροκατασκευαστική, έγιναν δεκτές οι προτάσεις αυτές από τους επιτρόπους τα Γιάννη Κρούς και ε, Γκέγαν Κουίν. Γιατί επιλέξαμε αυτές τις τεχνολογίες, να σας το εξηγήσω αυτό σύντομα. Αυτές οι βασικές τεχνολογίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή κάποιων προϊόντων. Το κινητό σας τηλέφωνο, οι περισσότεροι από σας έχετε ένα μαζί σας σήμερα. Στο τηλέφωνο αυτό έχουμε προχωρημένα υλικά Έχουμε ηλεκτρονικά τρανζίστορς, έχουμε τεχνολογίες σε επίπεδο νανοτεχνολογίας, έχουμε φωτογραφική τεχνολογία για βίντεο, για εικόνες, έχουμε ακόμα και βιοτεχνολογικά στοιχεία για την ταυτοποίηση των κλήσεων κτλ. Αν δείτε σαν παράδειγμα αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε για τον έλεγχο της γρήπης των πουλερικών. Όλες αυτές οι τεχνολογίες παίζουν ρόλο και μπορούμε να χαρακτηρίσουμε με τον ίδιο τρόπο όλα τα προϊόντα φωτοβολταϊκά. Προχωρημένα υλικά, ηλεκτρονικά, φωτονική, γενικά κάθε προϊόν το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι συνδυασμός κάποιων βασικών τεχνολογιών. Ένα τελευταίο παράδειγμα είναι το αυτοκίνητο. Σε ένα αυτοκίνητο φυσικά έχουμε πάρα πολλά ηλεκτρονικά. Το 70% της αξίας των αυτοκινήτων είναι τα ηλεκτρονικά. Έχουμε βιοτεχνολογία σε σχέση με κάποια υλικά που χρησιμοποιούμε για τα ελαστικά. Έχουμε φωτογραφική ε, τεχνολογία στον τομέα των ηλεκτρονικών, των λαμπτήρων κτλ. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν την σημαντικές αλλαγές σε όλους τους τομείς αυτούς. Παίρνω ένα παράδειγμα εδώ, περνώντας από τις βασικές τεχνολογίες, τα προϊόντα και τις λύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία, σαν παράδειγμα στην βιομηχανία που αφορά τους λαμπτήρες, την ηλεκτρονική βιομηχανία και βλέπει ότι στην αρχή όλων των αλλαγών είναι οι λεγόμενες βασικές τεχνολογίες. Η Ευρώπη πρέπει να ελέγχει αυτές τις τεχνολογίες εφόσον θέλει να ελέγχει τα προϊόντα τα οποία θα δημιουργήσουν και τις θέσεις εργασίας στο μέλλον. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ας δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με την ανάλυση αυτή. Χαίρομαι καταρχάς να πω ότι η Ευρώπη παραμένει στον αγώνα για την ανάπτυξη αυτών των βασικών τεχνολογιών, σε αυτούς που είναι στο πίσω μέρος της Βλέπετε το φάκελο τους τομείς ε, όπου είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, των ε, διπλωμάτων ευαισθητεχνίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πράσινο είναι της Ασίας και το οριζόντιο κομμάτι είναι αυτό το οποίο έχει η Ευρώπη. Σε επίπεδο ευαισθητεχνιών λοιπόν η Ευρώπη είναι πάντα από τους πρώτους. Βλέπετε όμως την ταχύτατη άνοδο της Αυστρίας. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για την αντιγραφή τεχνολογιών, μιλάμε για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και νέων προτάσεων. Η Ευρώπη λοιπόν παραμένει στον αγώνα και σε επίπεδο ε, τεχνιών η Ευρώπη έχει κεντρικούς θα έλεγα παίκτες, παράγοντες. Αν πάρουμε τις ευρεσιτεχνίες σαν δίκτυ δυναμικού ευρεσιτεχνίας και καινοτομίας, να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Τρεις, τρεις τομείς, τρία παραδείγματα μόνο, που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Σαν παράδειγμα μπαταρίες, ισορρευτές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φωτοβολταϊκά και ό,τι έχει σχέση με τις ε, ε, ανανεώσιμες πηγές. Σας μιλήσουμε για τους ισορρευτές. Τα, προσπαθώ να τα πω σχετικά απλά. Τα τρίγωνα τα οποία βλέπετε αντιπροσωπεύουν το μερίδιο των τριών ομάδων των χωρών, δηλαδή Ηνωμένε Πολιτείε, Ευρώπη και Ασία, σε επίπεδο ευρεσιτεχνιών. Εδώ βλέπετε ότι η Ευρώπη έχει το 20% στις ευρεσιτεχνίες ή μάλλον η ΕΠΑ 20%, 35% η Ασία, 31% εμείς. Είμαστε περίπου στο ίδιο επίπεδο. Αν δείτε τους κύκλους, οι κύκλοι αντιπροσωπεύουν την κατασκευή και τις θέσεις εργασίας βέβαια. Κοιτάξτε στην Ασία, 87% της κατασκευής γίνεται στην Ασία, λαμβάνει χώρα στην Ασία. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας, 1% στις Ηνωμένε Πολιτείες και 0% 0% στην Ευρώπη. Σε επίπεδο παραγωγής ισορρευτών υψηλού επίπεδου. Λοιπόν, σας δείχνω τι γίνεται. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει αγώνας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, νέων ηλεκτρικών οχημάτων και αυτά είναι στοιχεία εμπιστευτικά από το γραφείο του Προέδρου της Ρενό Βλέπουμε ότι στην Ασία σαν παράδειγμα 3,3 δις ευρώ επενδύθηκαν και 2,5 ακριβώς, 2,5 δις ε, για τις μπαταρίες, για τους ισορρευτές. Στις Ηνωμένε Πολιτείε 9,1 δις, 4,5 περίπου για τις μπαταρίες. Και στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξοδεύει 100 εκατομμύρια σε αυτό τον τομέα. Πώς μπορούμε να παίξουμε εμεί σε επίπεδο βιομηχανία με αυτά τα χρήματα. Και βλέπετε μετά τι κάνουν οι υπόλοιπες χώρες, Γαλλία και Γερμανία. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει η κατάσταση εδώ. Ο πρόεδρος Ομπάμα στην, κατάσταση, στην ομιλία για την κατάσταση της χώρας τον Ιανουάριο είπε ότι το βασικό μήνυμα είναι ότι άλλαξαν οι κανόνες και έδωσε άδεια στην κυβέρνησή τους, στη διοίκηση και στις πολιτείες να κάνουν ό,τι χρειάζεται έτσι ώστε να ξανακερδίσουν τον αγώνα για το διάστημα σαν παράδειγμα. Και όχι μόνο προφανώς συγκεντρώνουν την προσοχή τους και στον τομέα της επένδυσης, στον τομέα της καινοτομίας, αλλά βλέπετε εδώ για τον ιδρυτή της Intel, ο οποίος λέει ότι θα προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε τα προϊόντα μας και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Λοιπόν, προσπαθούν οι Αμερικανοί να ξαναρχίσουν να κατασκευάσουν και στις Ηνωμένε Πολιτείε, προσπαθούν να προσελκύσουν ξένες ε, εταιρείε. Η BASF έχει δημιουργήσει το πιο προχωρημένο εργοστάσιο α, μπαταριών. Η Shaft έφυγε από τη Γαλλία για διάφορους λόγους και θα ξεκινήσει στις Ηνωμένε Πολιτείες νέο εργοστάσιο. Λόγω ακριβώς των επιδοτήσεων για τις ΣΑΦΤ, σαν παράδειγμα, βλέπετε 200 ε, εκατομμύρια για το εργοστάσιο, το 50% προέρχεται από μια επιδότηση του Υπουργείου Ενέργειας, ενώ στην Ευρώπη εμείς ε, δεν έχουμε να βοηθήσουμε τίποτα, σε τίποτα και ίσα ίσα θα υπάρξουν και περιορισμό το ίδιο και για την ΠΑΣΦ, 50 εκατομμύρια αξίζει το εργοστάσιο, 24% επιδότηση από το Υπουργείο Ενέργειας. Βλέπουμε ότι χάνουμε τους βασικούς τεχνολογικούς μας παίχτες από τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Κίνα. Ας ένα δεύτερο τώρα για τη βιομηχανική βιοτεχνολογία. Και εδώ βλέπετε τα τρίγωνα, τα ποσοστά ευρεσιτεχνίας. Ποιος ηγείται η Ευρώπη, 36%. 34 από τη ΣΥΠΑ και 33 από την Κίνα. Αν δείτε για την κατασκευή, για την παραγωγή των προϊόντων, 54% στη ΣΥΠΑ, 5% και μειούται συνέχεια για την Ευρώπη. Έχουμε μια πλήρη ε, διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην επιστήμη από τη μία και τη βιομηχανία από την άλλη. Θα βελτιωθεί η βιομηχανία, η κατάσταση αυτή. Η βραζιλιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε 18 δις ε, ε, δολάρια επένδυση στον τομέα της, ε, του, της εθανόλης και του ζαχαροκάλαμου. Ενώ είχαν επενδύσει αντίστοιχα 6 δις το 2010. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, μετά από τις οδηγίες και του Προέδρου Ομπάμα έχει ανταγωνιστική στάση επιθετικά και συγκεντρώνει τους ηγέτες και στην κατασκευή. Η εταιρεία Ineos Bio που χρησιμοποιεί επαναστατικές τεχνολογίες προσελκύθη από τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, για ένα εργοστάσιο 130 εκατομμυρίων δολαρίων και 50 εκατομμύρια τα πήρε από το ε, αντίστοιχο Υπουργείο των Ηνωμένων Πολιτειών και με δανειακές εγγυήσεις. Δεν υπήρχε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κάνει κάτι τέτοιο εδώ στην Ευρώπη. Βλέπουμε λοιπόν οι καλύτερες και πιο καινοτόμες εταιρείες προσελκύονται στον υπόλοιπο κόσμο. Και ένα τελευταίο παράδειγμα είναι τα φωτοβολταϊκά. Είναι εξαιρετικός ο τομέας αυτός γιατί η Ευρώπη έχει τη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο. Η Ευρώπη όπως βλέπετε έχει το 77% της αγοράς. Η αγορά είναι εδώ μαζί μας στην Ευρώπη. Στην εφημερίδα σήμερα έλεγε ότι υπήρχε μία φωτογραφία του, προέδρου, του δημάρχου μάλλον του Φίλισμποργκ από την Γερμανία ο οποίος ήταν μπροστά σε φωτοβολταϊκά πινάκια. Δεν ήταν γερμανικά προφανώς. Η αγορά είναι στην Ευρώπη όμως. Ας δούμε πώς βρίσκεται η ευαισθητεχνία. Η Ευρώπη έχει κατατεθειμένα το 34%, η ΕΠΑ 27% και η Κίνα 42%. Για την κατασκευή η αγορά όπως είπαμε είναι στην Ευρώπη. Έπρεπε να έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής γιατί όπως είπα 77% της αγοράς είναι στην Ευρώπη και εμείς καλύπτουμε μόνο το 13% με τη δική μας παραγωγή. Κάναμε μια ανάλυση δείχνοντας τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν θέλαμε να βγει σε εφημερίδες κάτι τέτοια. Βλέπουμε την κατάσταση από το 2001 μέχρι το 2004, 9 και 10 για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Βλέπετε τις σημαίες της εθνικότητας των διαφόρων επιχειρήσεων. Πριν 10 χρόνια είχαμε 6 από τις πρώτες 10 εταιρείες φωτοβολταϊκών. Το 2009 έχουμε μία μία μοναχική παρά το ότι έχουμε τη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, παρά ότι συνεχίζουμε να εμένουμε στα φωτοβολταϊκά, αλλά παρόλα αυτά τι γίνεται με όλες τις άλλες επιχειρήσεις. Οι αμερικανικές, είχαν μία το 2001, έχουν μία το 2010, οι ασιατικές τώρα, οι Ιάπωνες σαν παράδειγμα, οι Ιάπωνες είχαν τέσσερις το 2001, 2 το 2009 και 2 το 2010. Λοιπόν, ποιος πήρε όλες τις θέσεις αυτές, αν το δούμε προσεκτικά, θα δούμε ότι είναι η λαϊκή Κίνα. 8 από τις 10 πρώτες θέσεις στα φωτοβολταϊκά, στην κατασκευή φωτοβολταϊκών κυψελών, είναι φυσικά κινέζικες και προφανώς τον χρόνο, του χρόνου η κατάσταση θα είναι ακόμα πιο σαφής. Δεν είναι δύσκολη η διαδικασία, μας λείπει κλίμακα για να μειώσουμε την τιμή. Χρειάζονται λοιπόν δάνεια και εγγύσει για τα δάνεια. 21 δις σε δάνεια πήγανε από τις τράπεζες στις κινέζικες επιχειρήσεις. 21 δις από κυβερνητικές τράπεζες, κρατικές ε, τράπεζες δάνεια εκτός ε, μάλιστα επιτοκίων αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν μπορεί να δώσει τέτοιου είδους δάνεια. Και η κατάσταση χειροτερεύει συνέχεια. Η Deutsche Bank είπε ότι ε, η Κίνα έκανε συμφωνίες με τις επιχειρήσεις στον τομέα αυτός για πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Η Jinko Solar πήρε ένα δάνειο 7,6 δις Μία εταιρεία 7,6 δις. Βλέπουμε μια κατάσταση λοιπόν όπου η αγορά για τα φωτοβολταϊκά είναι ευρωπαϊκή. Έχουμε χώρες όπως η Γερμανία που προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές Έχουμε τεράστια κίνητρα, πολλές χώρες ξοδεύουν ε, δις για τα φωτοβολταϊκά και τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στην Κίνα γιατί εκεί φτιάχνονται τα προϊόντα, εκεί βρίσκονται οι θέσεις εργασίας. Έχουμε στην Ευρώπη αυτό που θα ονόμασα την κοιλάδα του θανάτου ανάμεσα στην γνώση και την αγορά. Ξοδεύουμε περισσότερο από άλλους και από την Ασία για τη βασική έρευνα. Μιλάμε πάρα πολύ για τη βασική έρευνα. Ξοδεύουμε αναλογικά και έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία για τις ευαισθητεχνίες, αλλά δεν τα κάνουμε αυτά θέσεις εργασίας. Προσπαθούμε να δούμε λοιπόν πώς θα καλύψουμε, θα φτιάξουμε μια γέφυρα πάνω από αυτή την κοιλάδα του θανάτου να σταματήσω λέγοντας το τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Μίλησα για τους λαμπτήρες και για το φωτισμό γενικότερα. Ξέρετε ότι έχουμε τη Philips, άλλες εταιρείες. Θα έπρεπε να είμαστε ισχυροί. Αλλά το ίδιο ισχύει και με όπως και στα φωτοβολταϊκά. Βλέπουμε ότι το κόκκινο είναι τα υλικά, πράσινο ηλεκτρονικά, συστατικά είναι το κίτρινο και συστήματα το ε, μπλε. Η Κίνα φυσικά εδώ τα παίρνει όλα. Υπάρχουν κίνητρα 50% από πλευράς του κράτους για αυτόν τον πολύ στρατηγικό τομέα. Υπάρχουν ακόμα περισσότερα κίνητρα και για την κατασκευή των προϊόντων και από πλευράς της ε, τόνωσης της ζήτησης η Κίνα έχει ένα πρόγραμμα που λέγεται LED Cities. Έχουν βρει 21 πόλεις για την εγκατάσταση ε, φωτισμού με LED ε, σε, όλες τις, ε, σε όλους τους δρόμους αυτών των πόλεων. Σαν παράδειγμα στην επαρχία του Wandong έδωσαν 90 εκατομμύρια για να επιδοτήσουν έτσι ώστε το 30% των λαμπτήρων στους δρόμους του φωτισμού του δημοτικού να είναι LED. Εμείς έχουμε εξοδέψει 10 εκατομμύρια για να ανταγωνιστούμε την Κίνα στον τομέα αυτό όταν το είπαμε αυτό έτρεπαν οι Κινέζοι. Η κατάσταση δεν πάει καθόλου καλά λοιπόν σε άλλους τομείς όπου έχουμε ηγετική επιστημονική θέση, στις μαγνητικές μνήμες σαν παράδειγμα, που ξεκίνησαν και από την Γαλλία, από την Γκρενόμπλ, έχουμε την ηγετική όπως είπα επιστημονική γνώση Έχουμε πάρα πολλούς επιστήμονες που εργάζονται και βελτιώνουν. Έχουν δημιουργηθεί νέες επιχειρήσεις όπως η εταιρεία Κρόκους. Αλλά η εταιρεία αυτή δεν θα μπορούσε να βρει την κατάλληλη χρηματοδότηση και την δανειακή στήριξη. Και γι' αυτό λοιπόν αγοράστηκε για 300 εκατομμύρια από την Ρουσνάνο στη Ρωσία και φυσικά θα ξεκινήσει η παραγωγή των προϊόντων στην Ρωσία, ό,τι και με τα βολταϊκά, ό,τι και με τις μπαταρίες. Στις Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχει μια επιτροπή, το Προεδρικό Συμβούλιο για γνωμοδοτήσεις στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Δημοσίευσαν την παρούσα έκθεσή τους, λένε τα ίδια που λέμε και εμείς. Πρώτον λέγουν ότι θα πρέπει να ξεπεράσουν και αυτή αυτή την κοιλάδα του θανάτου μιλούν για να, την δημιουργία της υποδομής τεχνολογίας, όχι επιστήμης αλλά τεχνολογίας. Εμείς μιλάμε για επιστημονικές υποδομές αλλά δεν μιλάμε για τεχνολογικές υποδομές. Απαιτείται η επιτάχυνση της διαδικασίας κατασκευής και παραγωγής, θα πρέπει να υπάρξει συνδυασμός των κατασκευαστικών δυνατοτήτων και της έρευνας και της ανάπτυξης που συνδυάζεται με τις κατασκευαστικές δυνατότητες και χρειάζεται επίσης να δημιουργήσουν αυτό το οποίο ονομάζουν μια νέα πολιτική πρωτοβουλία για να καλυφθούν οι αδυναμίες της αγοράς σε σχέση με την Κίνα σήμερα. Εμείς είμαστε σε συζητήσεις με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Στις 28 Σεπτεμβρίου θα συναντηθούμε με τον Αλμούνια, αλλά μέχρι τώρα δεν κάναμε και πολλά πράγματα για να διευκολύνουμε την κατάσταση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ΣΥΠΑ και στην Ασία. Η Κίνα έχει βάλει τις αυτές τις επιχειρήσεις βασικής τεχνολογίας στο κέντρο της στρατηγικής τους. 18 από τις 100 ε, τόσες πρωτοβουλίες βασίζονται στις λεγόμενες βασικές τεχνολογίες. Δεν αναπτύσσουν μόνο τις δυνατότητες κατασκευής αλλά και τις τεχνολογίες. Κάναμε μια σύγκριση διεθνή σε σχέση με τα ποσοστά εφαρμοσμένων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από Κίνα, Κορέα κτλ. Πράσινο βλέπετε το ποσοστό της βασικής έρευνας. Βλέπετε τα ποσοστά για την Κίνα, την Κορέα και τη ΣΥΠΑ. 11% βασική έρευνα στην Κίνα, 24% στην Κορέα, αλλά 11% μόνο στην Κίνα, 32% στην Κίνα στην εφαρμοσμένη έρευνα και το 58% στην έρευνα για την ανάπτυξη, για την κατασκευή των προϊόντων. Στην Κορέα το ποσοστό είναι περίπου το ίδιο με τη ΣΥΠΑ, 24% βασική έρευνα, 32 με 28% εφαρμοσμένη έρευνα και αναπτυγμένη έρευνα 45% βλέπουμε ότι ο μέσος όρος είναι 25% βασική, 25% εφαρμοσμένη και ε, το υπόλοιπο 50% κατασκευή. Τι κάνει η Ευρώπη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοιχεία δεν έχουμε, δεν έχουν στόχους, δεν τους μετράνε. Έχουμε τα στοιχεία από τα κράτη-μέλη, προσθέτουμε βλέπετε τα στοιχεία, 36% βασική έρευνα, γιατί θέλουμε να έχουμε πολλές δημοσιεύσεις και ευαισθητεχνίες. Η πλευρά της χρηματοδότησης μυστήριο. Δεν μπορεί κανείς να αναλύσει τα στοιχεία, δεν μπορούμε να το δούμε. Με τον ίδιο τρόπο υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε, βλέπουμε πάντως πως έχει η κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας όχι μόνο στη βασική έρευνα, αλλά και στην αναπτυγμένη έρευνα και στην έρευνα ακριβώς την εφαρμοσμένη και πέραν της εφαρμοσμένης για τα πρωτότυπα που θα οδηγήσουν στην κατασκευή των προϊόντων εδώ. Αυτά είναι τα στοιχεία. Είναι πρώτη φορά που σας δείχνουμε τα στοιχεία αυτά και θα ζητήσω από οποιονδήποτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μου πει τι στόχους έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων και για τη βασική έρευνα και για την αναπτυγμένη έρευνα. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι οι συστάσεις από την ομάδα μας περιλαμβάνονται λεπτομερώς στην έκθεση που έχετε μπροστά σας. Υπογραμμίζω τρεις βασικές συστάσεις. Πρώτον, θα πρέπει αυτά τα ΚΕΤ να είναι βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη. Δεύτερον, ότι θα πρέπει η Ευρώπη να χρηματοδοτεί την έρευνα στο σύνολό της, όχι μόνο βασική έρευνα, αλλά και αναπτυξιακή έρευνα και έρευνα στον τομέα της κατασκευής. Δεν το κάνουμε αυτό. Εμείς μόνο το μπλε κομμάτι χρηματοδοτούμε. Βασική μόνο τεχνολογική έρευνα. 5, 6, 7, 8 δεν χρηματοδοτούνται στην Ευρώπη για διάφορους λόγους. Γιατί είμαστε υποτίθεται κοντά στην αγορά. Αλλά αυτό ε, δεν συμβαίνει στη ΣΥΠΑ και στην Ασία. Και τέλος, χρειάζεται να αλλάξουμε τους ορισμούς της έρευνας και της ανάπτυξης. Για να το κάνουμε αυτό χρειάζεται να αποκαταστήσουμε τις ισορροπίες των ερευνητικών προγραμμάτων και της καινοτομίας προτείνω να περάσουμε στις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθεί ο υπόλοιπος κόσμος. Αν η ΕΠΑ ξοδεύει μόνο 25% στη βασική έρευνα και η Κορέα το ίδιο, γιατί εμείς πρέπει να ξοδεύουμε πολύ περισσότερο και να μην βάζουμε χρήματα και στην αναπτυγμένη έρευνα και στην έρευνα την εφαρμοσμένη έστω. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα θέλω να υπογραμμίσω, το ότι στις Ηνωμένε Πολιτείε, όταν παίρνει κανείς χρηματοδότηση από το αντίστοιχο Υπουργείο ή την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, πρέπει να εκμεταλλεύεται ε, τις δυνατότητες που δίνει η χρηματοδότηση αυτή πρώτα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Λογικό. Στην Ιαπωνία, στην Κορέα, δεν θα αναφερθώ στην Κίνα καθόλου αν χρηματοδοτήσει από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, αναμένεται να εκμεταλλευτείς ακριβώς τις γνώσεις σου στη χώρα σου. Στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπάρχει καμία τέτοια υποχρέωση. Λοιπόν, χρηματοδοτούμε εμείς πάρα πολύ έρευνα και σε τομέα των φωτοβολταϊκών, των συσσωρευτών και σε άλλους τομείς και η κατασκευή γίνεται αλλού και στην ουσία τις γνώσεις αυτές μέσω πανεπιστημίων, ερευνητικών Ινστιτούτων, μέσω επιχειρήσεων τις στέλνουμε στο εξωτερικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν σε συνεργασία και με τον Επίτροπο Μισελ Μπαρνιέ και τον Επίτροπο Ταγιάννη να προσπαθήσουμε να έχουμε αναπτυγμένη έρευνα στην Ευρώπη, πραγματικά ευρωπαϊκή, ανταγωνιστική, όπως και στην Ασία ε, και τη ΣΥΠΑ. Ακούγεται απλά λογικό αυτό τα 56 δις αυτά τα οποία θα ξοδέψουμε στην περίοδο από το 2014 και μετά ή μέχρι 80 δις θα ξοδέψουμε για την καινοτομία και την έρευνα δεν υπάρχουν εγγυήσει ότι θα εκμεταλλευτούμε τα χρήματα αυτά κυρίως στην Ευρώπη. Περίεργο πράγμα. Δεν θα πρέπει όμως να το κάνουμε. Τέλος. Θα πρέπει να συνδυάσουμε τα διάφορα κοινωτικά προγράμματα. Ακούγεται απλό, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει σήμερα. Και τέλος, για τις κρατικές επιδοτήσεις. Ζητάμε εμείς να υπάρχει μια ρήτρα αντιστήχησης η οποία θα επιτρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου είναι στρατηγικά απαραίτητο να δίδει τα ίδια κίνητρα που δίνουν οι ανταγωνιστές μας στον κόσμο. Βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται η ΕΠΑ, πώς προσελκύει τους νεότερους και αποδοτικότερους επιστήμονες η Γενική Διεύθυνση ε, Καινοτομίας δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Έχουμε επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, συνδυάζει την επιστήμη, βλέπετε τα αποτελέσματα πολύ καλά στην επιστήμη, ηγέτες στον κόσμο στην επιστήμη την καθαρή. Αν ξοδεύαμε τα ίδια λεφτά και για την τεχνολογία, χρηματοδοτώντας, χρηματοδοτώντας την τεχνολογία, τους μηχανικούς, Όλα αυτά τότε θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις. Έχω 4.000 μηχανολόγους στον τομέα, σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Έχουμε ένα δάνειο μόνο που δίδεται, ένα ταμείο που δίδεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο α, Έρευνας Υπάρχουν πολλοί τομείς εξωτικοί που προκαλούν ενδιαφέρον και ζητούν χρηματοδότηση. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Τελειώνοντας, να κάνω τρεις βασικές προτάσεις για το πόσο ο πρόεδρος σας και εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε. Τα λέω ξερά, αλλά είναι μια ευκαιρία εδώ. Θα ήθελα να σας ζητήσω να βοηθήσετε να συστήσετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεσή μας, στις συστάσεων για τα ΚΕΤ. Η σωστή εκμετάλλευση δηλαδή των τεχνολογιών των ηλεκτρονικών στην Ευρώπη κτλ το να έχουμε ένα υπροπολογισμό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λέει θα ξοδέψουμε τόσα χρήματα για τη βασική έρευνα, τόσα για την αναπτυγμένη έρευνα και τόσα για την εφαρμοσμένη, αυτά όλα θα πρέπει να γίνονται στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας ζητήσω λοιπόν την βοήθειά σας να συστήσετε και εσείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει τις προτάσεις μας. Δεύτερον, θα ήθελα να ζητήσουμε ξεκάθαρους στόχους χωρίς αμφιβολίες στον τομέα της καινοτομίας και της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον προϋπολογισμό και για τη βασική. Και τέλος θα ήθελα να ζητήσω από σας Πρόεδρε να μας πείτε πως τους επόμενους μήνες μπορείτε να οργανώσετε μια μεγάλη ακρόαση για τα ε, εμπόδια στη λειτουργία των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα ΚΕΤ στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Νομίζω ότι η σημασία που έχει ο τομέας αυτός και οι θέσεις απασχόλησης, καλοπληρωμένων θέσεων απασχόλησης έχει μεγάλη σημασία και κάτι πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Green. Äh, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ εντυπωσιακή και πλούσια η παρουσίασή σας. Να, παρουσιάσω, να περάσουμε στην συζήτηση. Η κυρία Γκροστέτα έχει πρώτη το λόγο. Σας ευχαριστώ. Και θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμότατα για την παρουσίαση που μας κάνατε και που δυστυχώς δεν μας δίνει λόγο για αισιοδοξία γιατί ήσταν η απτή απόδειξη ε, μιας Ευρώπης ε, που μένει όλο και πιο πίσω και είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας υποβάλει πρόταση μέχρι το 2012 και όλους αυτούς τους μήνες σωρεύουμε τις καθυστερήσεις και χάνουμε όλο και περισσότερες θέσεις απασχόλησης όπως μας είπατε. Μας ε, παρουσιάσετε πολύ σαφώς τα πράγματα και πραγματικά ενισχύεται τα επιχειρήματα στην έκθεση που υπερψηφίσαμε πριν από λίγους μήνες για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική. Ήμουν σκιώδης συγγετρία της ομάδας μου για την Ευρωπαϊκή αυτή βιομηχανική πολιτική και πολλά τα στοιχεία που μας δώσατε ήδη τα είχαμε περιλάβει στην έκθεση αυτή με λιγότερο επίπεδο ακρίβειας βέβαια. Σίγουρα εσείς επιμείνατε σε πολλά επιμέρους σημεία και αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τους κανόνες μας γιατί αν δεν τους αλλάξουμε, τους κανόνες αγοράς και ανταγωνισμού, τότε δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα μας μιλήσατε για ακρόαση. Φυσικά χρειαζόμαστε ακρόαση, μια δημόσια ακρόαση στην οποία θα προσκαλούμε τους συναδέλφους που εργάζονται στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Ανταγωνισμού, γιατί η Επιτροπή Βιομηχανίας και Έρευνας είναι απόλυτα πεπισμένη για το όρθο των λόγων σας και συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Η έκθεσή μας για τη βιομηχανική πολιτική που κατατήθηκε από συνάδελφο της Σοσιαλιστικής Ομάδας, η έκθεση αυτή ε, εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Στην Επιτροπή μας υπήρχε ε, συνένεση, αλλά θέλουμε τη συμφωνία και των άλλων συναδέλφων που εργάζονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θα πρέπει και αυτούς να προσκαλέσουμε λοιπόν στη δημόσια κρόαση για να έχουν την ευκαιρία να σας ακούσουν. Μιλήσατε για την έρευνα. Φοβάστε ακόμη αυτό το φαινόμενο της διαφυγής των εγκεφάλων. Γνωρίζουμε ότι η ανώτατη εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια μας δεν είναι ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά συνεχίζεται αυτό το φαινόμενο της διαρροής, της διαφυγής των εγκεφάλων. Ή προσελκύουμε και εμείς ειδικευμένους ερευνητές από το εξωτερικό. Επίσης, πώς εξασφαλίσουμε καλή επικοινωνία ώστε να αποφύγουμε την ε, ε, δυσπιστία του πληθυσμού. Όταν μιλούμε για νανοτεχνολογία, ακόμη και στην Επιτροπή του Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαπιστώνουμε τεράστια δυσπιστία και επιφυλάξεις. Ο κόσμος φοβάται και οι συνάδελφοι ακόμη φοβούνται. Φυσικά είναι εύλογο να έχει κανείς προβληματισμό και όλοι μεριμνούμε για το περιβάλλον και την υγεία των συμπολιτών μας. Αλλά θέλουμε να προοδεύσουμε, θα πρέπει να βελτιώσουμε την επικοινωνιακή μας πολιτική και να εξηγήσουμε τα ωφέλη αυτών των νέων τεχνολογιών, που είναι πραγματικά τεχνολογίες καινοτόμες. Και τέλος, ε, κάτι που επίσης είχαμε αναφέρει στην έκθεσή μας για τη βιομηχανική πολιτική, θα πρέπει να πείσουμε ε, για την ανάγκη στους ε, κανόνες για το περιβάλλον και τους κοινωνικούς κανόνες ε, σε αυτή την τεράστια παγκόσμια αγορά να λάβουμε υπόψη και αυτό το Συμβούλιο για να αποφύγουμε τις καταστάσεις να τροποποιήσουμε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, να τροποποιήσουμε τους κανόνες για τη δημιουργία των σημαντικών ε, πρωταθλητών στην ευρωπαϊκή βιομηχανία για να μην μείνουμε πίσω ε, εξαιτία ε, του παροχημένου χαρακτήρα των κανόνων μας, που δεν προσαρμόζονται πια στην σύγχρονη πραγματικότητα. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση και η περιγραφή που μας κάνατε, αλλά εμένα πραγματικά με φοβίζει, με τρομοκρατεί θα έλεγα, γιατί μας δώσε την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοφεύει. Ότι αδιαφορεί πλήρως για τα επιχείρηματά σας και αυτό πραγματικά είναι πολύ ανησυχητικό. Έχετε επαφές ε, με τα κράτη-μέλη, με τους εκπροσώπους τους στο Συμβούλιο για παράδειγμα, ώστε να παρατηρήσουμε και το Συμβούλιο να προοδεύσει. Βέβαια, εν μέσω οικονομικής κρίσης είναι πολύ δύσκολο και στο συγγνώμη που μακρηγορώ, αλλά μας δώσατε απαντήσεις ε, για να διαφυλάξουμε και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης ακριβώς εν μέσω της κρίσης. Η κυρία Μαντουρέλ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ εκ μέρους της ομάδας μου να ευχαριστήσω ε, την παρουσία του Πρόεδρου της Ομάδας Εμπειρογνωμών Υψηλού Επιπέδου για την καταπληκτική παρουσίαση που μας έκανε και να συγχαρώ και ολόκληρη την ομάδα εμπειρογνωμόνων για το αξιόλογο έργο της. Συμφωνούμε με τα σχόλια, την ανάλυση, ε, τις προτάσεις σας και πραγματικά θα λαμβάνουμε δεόντως υπόψη τα μηνύματα αυτά και θα τα διαβιβάσουμε εκεί που χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους σημεία της έκθεσης, θα ήθελα να επισημάνω δύο που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικά. Δύο θέματα για τα οποία θα ήθελα τη γνώμη σας καταρχήν ό,τι αφορά το, τη δημιουργία του δυναμικού, των δυνατοτήτων και πώς ε, θα δώσουμε τέρμα σε αυτή την απομάκρυση, την αποσύνδεση της αγοράς από τα πανεπιστήμια, των επιχειρήσεων από τον ακαδημαϊκό κόσμο. Επίσης το θέμα της, του πολυδιάστατου χαρακτήρα, του πολυκλαδικού χαρακτήρα, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Όταν μιλούμε για τέτοιο διατομιακό χαρακτήρα. Τα θέματα αυτά τα εξετάσαμε και στα πλέσματα του 7ου ερευνητικού πλαισίου και μάλιστα οι τροπολογίες μας εγκρίθηκαν. Είπαμε ότι θέλουμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει διατομιακούς ε, κανονισμούς, αλλά διαπιστώσαμε ότι στην πράξη συνεχίστηκαν τα προβλήματα και οι επιφυλάξεις. Όχι τόσο από την Επιτροπή, όσο περισσότερο από την ε, επιστημονική κοινότητα. Από ό,τι κατάλαβα από την έκθεσή σας, ε, το βασικό πρόβλημα έγκυται στη δυσκολία που έχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεννοηθούν μεταξύ τους να καταλάβει ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να υπερκεράσουμε αυτά τα εμπόδια, πώς πιστεύετε ότι μπορέσουμε, θα μπορέσουμε να προωθήσουμε αποτελεσματικά αυτούς, τους πολυτομέα, αυτές τις πολυτομεακές προσεγγίσεις. Το θέμα αυτό της δημιουργίας δυνατοτήτων και δυναμικού με απασχολεί ιδιαίτερα. Τι νέες ειδικότητες, δεξιότητες, ή προγράμματα σπουδών πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε, τι μεταρρυθμίσεις ε, στον εκπαιδευτικό κλάδο ώστε να δημιουργήσουμε τέτοιο δυναμικό και να σταματήσει πια αυτή η απομόνωση, η αποσύνδεση του ακαδημαϊκού κόσμου των πανεπιστημίων από την αγορά και τι επιχείρησει. Ώστε γιατί πραγματικά για να δημιουργήσουμε τέτοιο δυναμικό και δυνατότητε, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό για να υλοποιήσουμε τους στόχους που μας αναφέρατε. Euh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κρίν, Κρέιν μάλλον, που μας έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση και παρουσίαση της έκθεσης, ε, πολύ επίκαιρη, γιατί εξετάζουμε τη μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική και το επόμενο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο. Έχουμε συζητήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με, με τις χώρες BRICS, με την Κίνα για το κλίμα και διαπιστώνουμε ότι αυτές οι μεγάλες χώρες του κόσμου που είναι ανταγωνιστές μας ε, για τους κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές ε, προσπαθούν να συμφωνήσουν μαζί, του, μαζί μας, αλλά προσπαθούν να πρωτοστατήσουν σε όλες τις μελλοντικές ε, πράσινες πολιτικές. Και ε, φαίνεται ότι μπορεί να υποβαθμίζουν, να υπονομεύουν σήμερα την διεθνή αλληλεγγύη, αλλά παρόλα αυτά κάνουν επενδύσει στη μελλοντική του ανταγωνιστικότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε εμεί την καλή στρατηγική, γιατί αν δεν επενδύσουμε εκεί που πρέπει και αν δεν έχουμε τη μέθοδο και ε, τα μέσα, δεν πρόκειται να κερδίσουμε ε, αυτήν την, ε, τον ανταγωνισμό, σε αυτόν τον ανταγωνισμό με τις υπόλοιπες χώρες. Αυτή η δύσκολη κατάσταση πρέπει να μας εξωθεί στο να λάβουμε ε, λύσεις, μέτρα. Οι συστάσεις είναι σύντομες και νομίζω ότι μπορούν να μας βοηθήσουν γιατί θα πρέπει πρώτα να διαμορφώσουμε μια συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να κινητοποιήσουμε όλες τις ομάδες γιατί οι τεχνολογίες αυτές είναι τεχνολογίες που συνδέονται με όλο το σύστημα παραγωγής. Είναι τεχνολογίες του μέλλοντος. Και θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις και να υποβάλω και κάποιες συστάσεις. Είπατε ότι σε ό,τι αφορά τους κανόνες του παιχνιδιού, φυσικά σε αυτή τη διαμόρφωσή του θα πρέπει να συμμετέχουν πολλές διευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να γίνει μια αναθεώρηση των κανόνων. Δεύτερο ζήτημα τη έκθεση. Τι αναπτυξιακή πολιτική που θα προτείνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα εφαρμόσουμε στα κράτη-μέλη θέλουμε. Θα θέλαμε η έκθεση αυτή να συνοδευτεί από χάρτες που θα εντοπίζουν τα σημεία που έχουμε ερευνητικές ομάδες, επιχειρήσεις, εκπαίδευση και ε, τα εργοστάσια για να δούμε πού βρίσκεται το δυναμικό και πώς θα το αξιοποιήσουμε. Έχουμε το πρόγραμμα Έρασμος. Γιατί να μην κάνουμε και εμείς όπως οι Αμερικανοί μια προσπάθεια εντοπισμού των νέων ερευνητών στα εργαστήρια και στο επόμενο πρόγραμμα να επενδύσουμε και στο θέμα αυτό. Σε μεγάλη κλίμακα, σε μεγαλύτερη από ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα γιατί έχοντα έτσι με Αμερικανούς που ασχολούνται με τα διπλώματα ευρεσιτεχνία στις ΗΠΑ, διαπιστώσαμε ότι αναζητούν ε, επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, αλλά τα διπλώματα ευρεσιτεχνία τα καταθέτουν και τα καταγράφουν στι ΗΠΑ. Παρόλο που οι εμπνευστέ του προέρχονται από διάφορα μέρη του κόσμου. Επίση, θα πρέπει να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μια δημοσιονομική μελέτη για να δούμε τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας ε, για να δώσουμε συνέχεια στις ερευνητικές προσπάθειες. Εγώ έκανα μια μικρή ανάλυση στην δική μου περιοχή και διαπιστώνω ότι στη Γαλλία ε, προσελκύουμε πολλές μικρές επιχειρήσεις ε, μεταφοράς ενέργειας χάρη στα φορολογικά κίνητρα που δίνουμε σε φορολογικές ελαφρύσεις για την έρευνα. Όταν όμως εξετάζουμε την αλυσίδα της καινοτομία και των αξιών, διαπιστώνουμε ότι δεν καταφέρουμε να προσελκύσουμε τους καλύτερους παραγωγούς. Χρειαζόμαστε ενισχύσεις και για τα καλύτερα προγράμματα και για την έμπρακτη εφαρμογή τους. Το ΛΙΤΕ είναι προσαρμοσμένο σε αυτά που το, οι, οι τεχνολογίες ε, ε, και πληροφορίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες μας για, την, ε, για τον εντοπισμό, προώθηση και υποστήριξη της πνευματικής ιδιοκτησίας. Θέλουμε στην ε, συζήτηση αυτή να συμπεριλάβουμε και τις επιχειρήσεις, ε, τον επιχειρηματικό κλάδο και τους επιστήμονες, γιατί υπάρχει το θέμα της συνολικής κινητοποίησης. Δεν θα πρέπει να κινητοποιήσουμε μεμονωμένα τους τομείς, αλλά όλους μαζί. Και μια ερώτηση που θα ήθελα να υποβάλω στον κύριο Κρέιν. Ήσταν αρκετά διακριτικός ό,τι αφορά τον αντίκτυπο τη έκθεση αυτής για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουμε συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ήθελε να συνδυάσει το πρόγραμμα πλαίσιο με τα προγράμματα καινοτομία. Ποια είναι η γνώμη σα, είναι σωστή αυτή η μέθοδο. ή μήπω ε, με βάση τα συμπεράσματά σα θα πρέπει να κάνουμε καλύτερη κατανομή των διαφόρων κονδυλίων των προγραμμάτων και την κατανομή τους ε, στα κράτη-μέλη σε σχέση με την υλοποίηση των στόχων τους. Ο κύριος Λάμπερτς. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κρίαν, εδώ βρίσκομαι. Προτού να προχωρήσω στον πυρήνα της παρέμβασής μου, θα ήθελα να θέσω μία συγκεκριμένη ερώτηση. Ε, τα ποσά που αναφέρατε είναι όλα ε, δημόσια κονδύλια, έτσι. Θα ήθελα να θέσω μία πρώτη ερώτηση. Ε, στη διαφορά ανάμεσα ε, στους ε, διαφόρους τομείς έρευνας. Βασική, ενδιάμεση κλπ. Αλλάζει η εικόνα, βλέπουμε τις του ιδίου τύπου διαφορές εδώ. Ωραία, ευχαριστώ. Και επίσης όσον αφορά την δημόσια συμμετοχή θα ήθελα να επικεντρώσω την παρέμβασή μου σε μια συγκεκριμένη πτυχή στα χρήματα. Δεν θα συζητήσω όλα τα νομοθετικά και ρυθμιστικά θέματα. Ε, θα αναφερθώ στα χρήματα γιατί δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το περιβάλλον μας. Δεν μας περισσεύουν τα χρήματα όπως περισσεύουν στην Κίνα. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, στην Κίνα ε, λαμβάνουν άφθονη χρηματοδότηση από το κράτος. Ε, εμείς ε, στο εγγύς μέλλον δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω να είμαστε σε θέση να δώσουμε εντολές στον τραπεζικό μας τομέα να χρηματοδοτήσει έρευνα και δεν έχουμε τα Δεν έχουμε τεράστια πλεονάσματα για να χρηματοδοτήσουμε τέτοια προγράμματα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε σοφή χρήση των χρημάτων που έχουμε στη διάθεσή μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι, όταν λέτε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα ε, για το τελευταίο κομμάτι της ε, εξίσωσης, ε, εσείς τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να διοχετεύσουμε χρήματα από την βασική έρευνα στην φυρμοσμένη έρευνα σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Αυτή είναι η πρώτη πτυχή. Ε, και δεύτερον, η ερώτηση... Η δεύτερη ερώτηση είναι ότι η Ευρώπη δεν έχει την δυνατότητα να... Ε, μάλλον η Ευρώπη δαπανεί χρήματα σε μεγάλα έργα. Ε, βρισκόμαστε καθοδόν να δαπανίσουμε 10-12 δισεκατομμύρια στο ίτερ. Μπορεί να σας αρέσει ή όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα και πάνω από 10 δισεκατομμύρια θα ε, χρησιμοποιήσουμε για το Γαλιλαίο. Το μήνυμα που ε, εξάγω από τα όσα μας είπατε είναι ότι βασικά δεν θα πρέπει να επενδύουμε σε αυτά ή θεωρείτε ότι και αυτά είναι ε, ε, βασικές ε, τεχνολογίες γενικής εφαρμογής. Το ίτερ μπορεί να μας δώσει αποτελέσματα ή όχι μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια, αλλά για το Γαλιλαίο έχω αμφιβολίες. Μπορεί τελικά να καταφέρουμε να προσωμιώσουμε τεχνολογίες ε, οι οποίες ήδη υπάρχουν και οι οποίες δεν ε, θα δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ευρώπη. Τα καλά νέα είναι ότι εσείς μπορείτε να κινητοποιήσετε μεγάλα προγράμματα, εφόσον είναι τα σωστά προγράμματα αυτά. Και πάλι δεν βρισκόμαστε σε θέση να συλλέξουμε τεράστια ποσά δημοσίου χρήματος. Τα μεγαλύτερα ποσά που μπορεί να επενδυθούν ε, στην Ευρώπη τα επόμενα δέκα ή περισσότερα χρόνια θα είναι ιδιωτικά ποσά. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αποφασίσουν ε, αν ε, θα πραγματοποιηθούν μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Όταν ακούω τους επιτρόπους που είναι αρμόδιοι για ε, ε, χρηματοοικονομικά θέματα και που μου λένε ότι αυτά είναι θέματα φορολογίας, αν ακολουθήσω τη δική τους ε, γραμμή σκέψης, τα χρήματα που θα είναι διαθέσιμα για τέτοιου τύπου δραστηριότητες, μάλλον προς τον νότο θα διοκετεύονται παρά προς τον βορρά. Ε, μ' αρέσει το αίσθημα του επίγοντος που έχετε. θα περίμενα Μ' αρέσει η ειλικρίνεια σας, ε, αλλά θα ήθελα εξίσου ειλικρινή απάντηση από εσά προ του πολιτικού σχετικά με τι επιλογέ που θα πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ. Ε, συνάδελφοι, ε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ε, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση. Ε, είναι ένα θέμα αποφασιστική σημασίας ε, για το μέλλον της Ευρώπης. Η πρώτη μου ερώτηση όταν μιλάμε για την τεχνολογία ε, λόγω της μικρής οθόνης ήταν δύσκολο να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση στις οθόνες αυτές εμείς που καθόμαστε εδώ πίσω. Μήπως θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε σε χαρτί την παρουσίαση αυτή. Τη δεύτερη μου ερώτηση την ανέφερε ήδη ο συνάδελφος Λάμπερτς. Ε, συμφωνώ μαζί του όσον αφορά τη χρηματοδότηση στην Ευρώπη, όσον αφορά το οικονομικό μοντέλο. Η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Και όσον αφορά τη λέξη κλειδί Κίνα, την πρόκληση της Κίνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα έχει ε, μεγάλες επιτυχίες όσον αφορά τις εξαγωγές, έχει ε, τεράστια κρατικά αποθέματα Τα κέρδη όμως ε, από αυτές τις ε, εξαγωγικές επιτυχίες ε, δεν θα τα απολαύσει ο λαός. Το θέμα είναι λοιπόν αν μπορούμε να αντιγράψουμε στο κινέζικο μοντέλο και αν είναι επιθυμητό στο κάτω-κάτω. Για μένα η απάντηση είναι απλή. Εδώ υπάρχει ένα κενό Ε, θα πρέπει να πάρουμε δημόσιο χρήμα και εάν πάρουμε δημόσιο χρήμα ε, έχει λυθεί το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο απλή απάντηση. Ε, και σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει σημαντική κρατική βοήθεια, παρόλα αυτά το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό. Γι' αυτό η ερώτησή μου είναι, σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείες, Στις Ηνωμένε Πολιτείε το δημόσιο χρήμα είναι που ε, δίνει τη δυνατότητα στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, για τις ε, παραγωγικές της επιτυχίες. η αιτία για το μεγαλύτερο παραγωγικό δυναμικό είναι το δημόσιο χρήμα. διότι στην πράξη τίθεται το ερώτημα εάν ε, τα διπλώματα ευρυστεχνίας από μόνα τους ε, είναι ο σωστός δείκτης. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφτηκα διάφορες μικρές επιχειρήσεις που μου έλεγαν ότι ε, δεν θέλουν να κάνουν αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διότι αφενός δεν θέλουν να δημοσιεύσουν τις τεχνολογίες τους και φοβούνται και το υψηλό κόστος. Μήπως ε, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Χέρτσογκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι και από την Ουγγαρία ε, προέρχομαι. Ε, μ' άρεσε πάρα πολύ η έκκλησή σας ε, να απλοποιήσουμε τα πράγματα. Κάποια θέματα θα ήθελα να θίξω. Πρώτον, ε, τα χρήματα. Ως ε, εισηγήτρια επί κάποια χρόνια για ε, τον προϋπολογισμό και για άλλα σχετικά θέματα, θα ήθελα να σας δώσω ένα ή δύο νούμερα. Είπατε ότι μία επιχείρηση στην Κίνα θα έχει κέρδος του χρόνου 7,6 δισεκατομμύρια, ε, ως, ε, όχι κέρδος, ε, συγγνώμη, ε, ως εγγύηση χρέους. το συνολικό, ο συνολικός περιπολογισμός του ε, προγράμματος πλαισίου 7 ανέρχεται επίσης σε 7,6 δισεκατομμύρια. 7,4 για τον ανταγωνισμό είναι ο προϋπολογισμός. Εσείς ε, στα 10 σημεία που αναφέρατε, αναφέρατε ε, διεύρυνση. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς τον προϋπολογισμό. Η απάντησή μας λοιπόν σε αυτό είναι περισσότερη Ευρώπη. Αλλιώς αν απλά διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή ε, χωρί να αυξήσουμε τον προπολογισμό, ε, σύντομα δεν θα έχουμε χρήματα για να τα πραγματοποιήσουμε αυτά. Δεύτερον, δεν αναφέρθηκε, θα ήθελα όμως να το αναφέρω. Εδώ και 7 χρόνια εγώ αγωνίζομαι για τις ε, βιομηχανίες ε, που αναφέρατε. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω την νομοθεσία, διότι θυμάμαι ότι ήμουν ασκιώδης εισηγήτρια για το REACH και την ε, ε, ε, και την επίδραση που θα έχει στις μπαταρίες. Εμένα, με ενδιαφέρει πολύ το θέμα των μπαταριών. Πολλά παιχνίδια έχουν μέσα μπαταρίες. Ακόμα και κούκλες τύπου Barbie έχουν μπαταρίες μέσα μερικές φορές. Η νομοθετική μας ισχύς για τις, όσον αφορά τις βιομηχανίες αυτές είναι τεράστια το 2005 είχαμε το ίδιο για, τον φωτισμό και τη βιοθανόλη. Και πέρσι είχαμε ακριβώς ε, το ίδιο για τα διανοητικά δικαιώματα, τα IPR. Η καλύτερη νομοθεσία, ε, πιστεύω λοιπόν ότι είναι θέμα κλειδί, δεν το αναφέρατε, αλλά νομίζω ότι είναι προφανές. Και δεν θα πρέπει να είναι μόνο καλή νομοθεσία, θα πρέπει να είναι και απλή, διότι όταν μιλάμε για έρευνα, μιλάμε για θέματα πολύ ελκυστικά. Εσείς αναφερθήκατε σε πολύ βασικές βιομηχανίες, ε, τον φωτισμό, την ε, εθανόλη. Νομίζω ότι η εθανόλη είναι από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα. Η βιοεθανόλη μπορεί να μην ε, φαίνεται το πιο ενδιαφέρον θέμα στον κόσμο, αλλά μιλάμε για απλές βιομηχανίες και το τελευταίο μου θέμα είναι ε, ότι θα ήθελα να σας προτείνω να υποβάλλετε την παρουσίασή σας ε, στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού. Το πρόβλημά μας είναι ότι ε, εμείς αγωνιζόμαστε όχι με ομοτήμους αλλά με υπουργούς οικονομικών. Ε, το θέμα κολλάει στα χρήματα και όχι στα θέματα παραγωγής. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Διότι οι μέτοχοι μπορεί να βρίσκονται ε, πολύ μακριά από τις μετοχές τους, ε, αλλά η ε, παραγωγή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στα κεφάλαια. Συγγνώμη που έχω πολλές ερωτήσεις, ε, αλλά ε, αναφερθήκατε σε θέματα που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνική. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω θερμά κύριε Κρίν για την ε, παρουσίασή σας. Μας ανοίξετε τα μάτια. Αναφερθήκατε και στη δική σας πατρίδα και εκλογική περιφέρεια και εμείς έχουμε εμπειρίες από τη δική μας και χαιρόμαστε που έχουμε μια πολύ απτή και συγκεκριμένη έκθεση με ποσοτικά στοιχεία και αριθμητικά στοιχεία. Θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο καμπής και να τροποποιήσουμε πραγματικά τα πράγματα. Υποβάλλεται πολλές προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης και είναι πολύ εύστοχες αυτές οι συστάσεις. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Δεν υπάρχει ε, ηγετικός ρόλος ε, δυστυχώς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Αντιμετωπίζουμε κρίση και βλέπουμε τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε ε, και στον τομέα αυτό. Δεν υπάρχει πρόβλημα μόνο με την έλλειψη χρημάτων. Φυσικά χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Αλλά μια και δεν έχουμε αρκετά χρήματα, θα πρέπει να ταξινομήσουμε, να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες μας και εκεί είναι το πρόβλημα. Έτσι λειτουργεί η Ευρώπη, όπως είπε ο κύριος Λάμπερτ θα πρέπει να ικανοποιήσουμε έστω και λίγο τους πάντες και ο καθένας έχει τα, τις δικές του προτεραιότητες. Θα πρέπει να επενδύσουμε φυσικά περισσότερες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και να τις θέσουμε ως μεγάλη, σημαντική προτεραιότητα. Δεύτερον, το θέμα δεν είναι περισσότερα κονδύλια, αλλά τα κονδύλια που έχουμε όχι μόνο για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και για το επόμενο βήμα να αξιοποιηθούν δεόντως. Και εκεί μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας. Δυστυχώς είναι ενησυχητική αυτή η έλλειψη στοιχείων αριθμητικών και θα πρέπει να επισημάνουμε αυτό το έλλειμμα. Κύριε Κρέιν, ε, δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η μόνη λόγη ε, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα ε, είναι μερικά από τα αίτια του κακού, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες αιτίες για αυτή την καθυστέρηση, την υστέρησή μας. Θα πρέπει να ελέγξουμε την κατάσταση και στα κρατη Φυσικά υπάρχουν διαφορέ μεταξύ του, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα είδο ε, γενική συνοτροπία και κουλτούρα στα κράτη-μέλη που αναχαιτίζει την πρόοδο ή δημιουργεί εμπόδια στην πρόοδο. Αν αποφασίσει κανεί να κατασκευάσει ένα νέο εργοστάσιο ε, και να συμπεριλάβει, να προωθήσει αυτές τις τεχνολογίες ε, στην αγορά, στην Κορέα μέσα σε έξι μήνες θα μπορεί να το κατασκευάσει και στην Ευρώπη δεν θα έχει περάσει ακόμη από τη φάση της άδεια μέσα σε ένα εξάμεινο. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, ώστε και στα κράτη-μέλη, στις πατρίδες μας, να δημιουργήσουμε εργαστήρια, όχι μόνο για τις τεχνολογίες, αλλά για τον τρόπο χορήγησης αδειών και για την επιτάχυση των διαδικασιών. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το επεξεργαστούμε περαιτέρω. Και κάτι άλλο, δεν υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία, αλλά ήδη αυτά που μας δώσετε μας δίνουν βασικές δείξεις. Εμείς ε, θα μπορούσαμε από κοινού με τις ΗΠΑ και τις άλλες ηγετικές δυνάμεις ε, να εξασφαλίσουμε όχι μόνο τις τεχνολογίες αλλά και τις βιομηχανίες. Και δυστυχώς δεν έχουμε πια το ανθρώπινο δυναμικό που χρειαζόμαστε. Και φαίνεται ότι φοβόμαστε να διακινδυνεύσουμε. Και αυτό φυσικά έχει κάποια σχέση με, τη, με τους χαλεπούς καιρούς και την κρίση που διανύουμε, αλλά και με το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Όχι ε, από τα πανεπιστήμια, αλλά από την στοιχειώδη εκπαίδευση. Μακροπρόθεσμα και αυτή η αναθεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος θα πρέπει να ενταχθεί στους στόχους μας. Ευχαριστώ κυρία Τόγια. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας. Μας έκανε πράγματι εντύπωση. Εσείς ουσιαστικά με συγκεκριμένα δεδομένα και με πολύ πιστικό τρόπο ε, μας δείξατε μια κατάσταση που όλοι κατανοούμε βέβαια και βλέπουμε τη σύγκριση θα έλεγα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου. Και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω από τον Πρόεδρο και τους συντονιστές να μελετήσουμε λίγο το θέμα αυτό για να δούμε αν μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα σημαντικά τα οποία ακούσαμε, με ποιους να μιλήσουμε, να ξεκινήσουμε μια συζήτηση με τις άλλες επιτροπές και να εμβαθύνουμε στο θέμα Είναι σαφές ότι τέτοιου είδους φαινόμενα και τέτοιου είδους εξελίξεις μας δείχνουν ότι η Ευρώπη τελικά είναι ακατάλληλη πλέον σε ορισμένους τομείς και πολιτικά. Απαιτείται να υπάρξει ένα νέο όραμα, μια μεγάλη αναπτυξιακή κοινοτική πολιτική, όχι μικρά επιμέρους μέτρα, και μέσω συγκεκριμένων βιομηχανικών πολιτικών, μέσω του προϋπολογισμού, μέσω του ανταγωνισμού, μέσω της έρευνας να μπορέσει να ανακτήσει τη δυνατότητα η Ευρώπη <clears throat> να σταθεί στο ύψος αυτών των οραμάτων και των στρατηγικών πολιτικών που απαιτεί η καθημερινότητα, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο κρίσης. Το πρόγραμμα λοιπόν είναι τεράστιο και θα πρέπει λοιπόν να μας βοηθήσετε να ασχοληθούμε με πιο συγκεκριμένα θέματα. Υπάρχει μία συνάδελφος η οποία ασχολείται ειδικότερα με τον προϋπολογισμό και γνωρίζει το τι πόρους δίνουμε σε σχέση με τον τομέα που μας ενδιαφέρει. Είναι περιορισμένοι πόροι οι οποίοι όμως θα έλεγα επιτρέπω να υπάρξει μια κάποια σύγκληση και θα πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε καλύτερα. Εγώ δεν κατάλαβα αν τα επιπλέον προγράμματα που προβλέπουν την συγχρηματοδότηση θα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν ή θα πρέπει κάθε χώρα να υπερασπίζεται τα δικά της προγράμματα. Πώς μπορούμε λοιπόν να συνδυάσουμε καλύτερα αυτού του είδους τα προγράμματα, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα ξεχωριστά κεφάλαια της ευρωπαϊκής πολιτικής. Έχουμε τα διαφορετικά ταμεία από τη μία. Κάποια από αυτά βοηθούν με έμεσο τρόπο και την έρευνα και την ανάπτυξη Θα πρέπει να προσπαθήσουμε βέβαια να συνοδεύσουμε αυτές ε, τις ρυθμίσεις με, συγκεκριμένες, ε, με συγκεκριμένους κανόνες. Γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι δεν θα προχωρήσουμε. Το πέρασμα από την ευαισθητεχνία στο πιλωτικό πρόγραμμα και τελικά στην παραγωγή απαιτεί πάρα πολύ ε, χρηματοδότηση ενδιάμεση. Υπάρχει μια σειρά λοιπόν επιμέρους μέτρων τα οποία θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα της πίστοσης, της απλούστευσης των διαδικασιών και του τι θα ακολουθήσει, ποια θα είναι η συνέχεια στην ευαισθητεχνία. γιατί πάρα πολλά μένουν σε επίπεδο δημοσιεύσεων και ευαισθητεχνιών μόνο και δεν πίνονται στις βιβλιοθήκες και δεν προχωρούν περαιτέρω. Τι κανόνες λοιπόν διαδικαστικούς, λειτουργικούς, φορολογικούς μπορούμε να θεσπίσουμε για να προχωρήσουμε. Κάθε χώρα να προσπαθήσει να είναι πιο ελκυστική από μόνη της μέσω κάποιων ρυθμίσεων φορολογικών εθνικών. Δεν νομίζω ότι η Ευρώπη στα πλαίσια της παγκόσμιας πρόκλησης θα πρέπει να επιλέξει τον δρόμο της του εσωτερικού ανταγωνισμού. δική μου χώρα ούτε καν αυτό δεν προσπαθεί να κάνει. Ή μήπως θα πρέπει όλη η Ευρώπη μαζί να βρει μια κάποια κοινή αντίληψη για τα πράγματα Ένα τελευταίο ερώτημα έχει σχέση με το λειτουργικό κομμάτι της δουλειάς μας. Έχουμε και εμείς ένα Ινστιτούτο λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Τεχνολογιών, που κάνει πιστικές όπως είπα παρουσιάσεις και ακολουθεί τον σωστό δρόμο από ό,τι φαίνεται. Πώς συνδυάζεστε μαζί τους. Εσείς προτείνετε επίσης και ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνολογίας πέραν της έρευνας ένας οργανισμός επιπλέον. Αυτό με ενοχλεί. Γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει αυτός ο οργανισμός, τι έχει να προσφέρει. Θα είναι στοιχείο αποτελεσματικότητας ή στοιχείο περαιτέρω υποδιαιρέσεων των λίγων πιστώσεων που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ. Ακούσαμε διάφορες ερωτήσεις. Ε, να προσθέσω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση του κύριου Κρέαν. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο ερώτημα γιατί πετυχαίνουμε γιατί δεν πετυχαίνουμε όλα αυτά που έχουμε να τα μετατρέψουμε σε ε, παραγωγικό πλεονέκτημα. Ε, φταίει η χρηματοδότηση, φταίνε οι πολύπλοκες διαδικασίες ή μήπως φταίει ότι οι ε, πολιτικές μας αποφάσεις δυσκολεύουν τη ζωή όσων θέλουν να προχωρήσουν στην παραγωγή. Ε, διότι εάν ισχύει αυτό τότε είναι ευθύνη δική μας και θα πρέπει εμείς ε, να ε, αντιδράσουμε διαφορετικά. Μήπως εμείς με την ομοθεσία μας δυσκολεύουμε τα πράγματα στην Ευρώπη, ίσως να το κάναμε θελημένα και να άξιζε τον κόπο, αλλά τότε δεν θα πρέπει να παραπονιόμαστε. Εάν όμως δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μας, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως θα πρέπει να επανεξετάσουμε τα νομοθετικά μας μέτρα. Είναι μια συζήτηση που έχουμε συχνά όταν μιλάμε για την νομοθεσία. Θα πρέπει να μιλάμε για τον αντίκτυπό τη. Θα πρέπει να βλέπουμε αν το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στην πρόθεσή μας. Πιστεύω ότι όταν ε, ανοίγει κανείς τη συζήτηση αυτή θα πρέπει να την ε, συνεχίσει μέχρι το τέλος. Χρήσιμο θα είναι να έχουμε μια αίσθηση ε, πόσο μεγάλο ποσοστό των προβλημάτων έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση, πόσο έχει να κάνει με τις διαδικασίες και πόσο έχει να κάνει με την νομοθεσία. Πόσα. Κύριε Κριέν. Κριέν. Ακούσαμε πολλές ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας δώσω την ευκαιρία να απαντήσετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους όσους υπέβαλαν ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω με τη σειρά. Κυρία Γκροστέτ, στα γαλλικά, ε, θερμά ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Επαφές με τα κράτη-μέλη. Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω ότι τρία από τα κράτη-μέλη, η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και οι υπουργοί τους, η Edith Cresson από τη Γαλλία, ο Υπουργός Παιδείας στην Μεγάλη Βρετανία και ο ομόλογος από τη Γερμανία, συνέταξαν κοινή επιστολή αμέσως μετά την έκθεση, τη συνυπέγραψαν εκφράζοντας την αμέριστη υποστήριξή τους προς τις συστάσεις της έκθεσής μας. Αυτή την επιστολή μπορούμε να σας την ε, διαβάσουμε μέσω της γραμματείας σας και να την ε, μελετήσετε. Περιμένουμε αντίστοιχε επιστολές από την Πολωνία και την Ισπανία. Υπήρξε κάποια καθυστέρηση λόγω των θερινών διακοπών. Οπότε Έχουμε ήδη εκδηλώσεις ε, ενθουσιώδους υποστήριξης από πολλά κράτη-μέλη και μάλιστα ε, ζήτησαν την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης οι χώρες αυτές. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν συγκεκριμένο κονδύλιο, συγκεκριμένη δημοσιονομική γραμμή για προγράμματα multicats, για προγράμματα που ε, εφαρμόζουν διαφορετικές βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής. Στην πράξη βέβαια και πολλοί το ανέφεραν. Ακριβώς εξαιτία του διατομιακού χαρακτήρα των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, γιατί σε ένα κοινικό χρειαζόμαστε και ηλεκτρονικά και φωτονικά, είναι εξορισμού ε, διατομιακές αυτές οι βασικές τεχνολογίες και έχουμε και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Πλαίσιο, αλλά εμπίπτουν ε, οι βασικές τεχνολογίες σε διαφορετικές γενικής διεύθυνσεις, ε, φωτονική και ηλεκτρονική σε μια γενική διεύθυνση και ε, και έτσι για υλικά και κατασκευή στην ε, Γενική Διεύθυνση Καινοτομία ε, και Έρευνα. Η βιοτεχνολογία εμπίπτει στι αρμοδιότητε άλλη Γενική Διεύθυνση. Βέβαια υπάρχει κατακαιρματισμό. Και απαντώντα στι επιστολέ των Υπουργών είπαμε ότι δυστυχώ ε, δεν έγινε μια σύζευξη των βασικών τεχνολογιών Εξαιτία του διατομιακού του χαρακτήρα. Πιστεύουν ότι θα πρέπει η φωτονική να παραμείνει στη γενική διεύθυνση και τα υλικά να εμπίπτουν στην, ε, σε άλλη γενική διεύθυνση έρευνα και Κοινοτομία. Βλέπετε τι προβλήματα όμω δημιουργεί αυτό ο κατακαιρματισμός. Πάντω προτείναμε μια ξεχωριστή δημοσιονομική γραμμή για τα Multicats και μάλιστα η Γενική Διεύθυνση Βιομηχανία ε, εξετάζει την πρόταση αυτή. Έχουμε την επόμενη εβδομάδα συνάντηση για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο εκπρόσωπο. Πάντως τα προγράμματα με μονομένες βασικέ τεχνολογίε ε, σε ξεχωριστέ διευθύνσει και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Θέλουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για πολλές ε, και συνδυασμένε βασικές τεχνολογίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε ε, έξι τέτοιες βασικές τεχνολογίες στην ομάδα εμπειρογνωμόνων. Μπορούμε να τις συνδυάσουμε, γιατί έτσι θα μπορούμε πραγματικά να κατασκευάσουμε διαφορετικά προϊόντα, να μην τρέχουμε από τη μια διέθεση στην άλλη. Φανταστείτε τι περίπλοκες θα είναι κοινέ προκηρύξεις διαγωνισμών, όταν πολλές ε, διευθύνσεις ε, εμπλέκονται. Η Samsung ήταν ανταγωνιστική Ακριβώ επειδή είχε συγκεντρωμένες όλες αυτές τις αρμοδιότητες για τα υλικά, για τι οθόνε, τα ηλεκτρονικά, το φωτενική, το λογισμικό, όλα σε, σε έναν ενίο φορέα. Γι' αυτό και προωθήθηκε στου στους διαγωνισμούς. Και εμεί ακριβώ εξαιτία του κατακαιρματισμού χάσαμε πολλέ θέσει απασχόληση. Υπάρχει θετική ανταπόκριση από τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να, να βρούμε ανταπόκριση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαφυγή εγκεφάλων. Όντω, στι ΗΠΑ οι εταιρείε ε, λαμβάνουν περισσότερη χρηματοδότηση και φυσικά μετακινούνται μαζί με το προσωπικό τους. Θέλουμε τους πιο ειδικευμένου εμπειρογνώμονες των τεχνολογιών και έχουμε πολλές ειδικευμένε ε, ε, τεχνολογίες για την επιστήμη. Και μάλιστα, πολλές φορές αν κανείς εξετάζει ένα σαλιγκάρι έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να λάβει χρηματοδότηση από ότι αν είναι σε μια καινοτόμα τεχνολογία διατομεακή, γιατί εκεί χρειάζονται πολύ περισσότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες, εμπλέκεται και ο ακαδημαϊκός κλάδος. Και εκεί έχουμε τεράστια προβλήματα. Αν δαπανούμε ένα ευρώ για την ε, επιστήμη θα πρέπει ένα ευρώ να το δαπανούμε και για την τεχνολογία, για την καινοτομία, ώστε τις ιδέες των πανεπιστημίων να τις μεταφέρουμε και να τις ε, πραγματοποιούμε στην αγορά. Θα πρέπει να έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για την τεχνολογία και όχι μόνο ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την επιστήμη όπως ισχύει τώρα. Θυμάμαι όταν ήμουν στην Ολλανδία δημιουργήσαμε ένα ε, Ιρλανδικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την τεχνολογία, την επιστήμη και τη μηχανολογία. Και αυτή ήταν η πρότασή μας και μάλιστα είχαμε διαπραγματεύσει με τον Ιρλανδό Υπουργό για μήνες ολόκληρους για να μην περιοριστούμε σε Συμβούλιο Επιστήμης μόνο, να περιλάβουμε και τις τεχνολογίες. Και νομίζω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Επιστήμη είναι πολύ περιορισμένο και δεν δίνει σωστή έμφαση. Θα πρέπει να μην δώσουμε έμφαση μόνο στην επιστήμη αλλά και στην τεχνολογία. Έχουμε λοιπόν επαφές με τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει αυτή να μεταφραστεί σε δράση έμπρακτη. Ίσως θα μπορούσατε ε, να έχετε επαφή με την Υπουργό Μπρέσον και άλλε για να δοθεί μια συνέχεια σε αυτή την επιστολή. Και να, για να σταματήσουμε τη διαφυγή των εγκεφάλων θα πρέπει και τα χρήματα που έχουμε να τα χρησιμοποιήσουμε πιο έξυπνα. Αυτό περισσότερο μας ενδιαφέρει, σωστή αξιοποίηση. Κύριε Μαδουρέλ, μιλήσατε για τη δημιουργία δυνατοτήτων δυναμικού και την αποσύνδεση πανεπιστημίων από την αγορά. Ε, ασχολήθηκα με πολλά startups, ήμουν καθηγητή και σε πανεπιστήμιο και νο, νομίζω ότι χρειαζόμαστε καλή οργάνωση στην καλύτερη οργάνωση στην Ευρώπη. Τα πανεπιστήμια πιστεύω ότι δεν είναι προγραμματισμένα, σχεδιασμένα για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, για να πάνε το α στο β. Έχουμε υποδομές, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε καλύτερη μετάβαση από, τη, από τα πανεπιστήμια στην αγορά. Έχουμε πολλές μεμονωμένες πρωτοβουλίες στη Γαλλία, στα, στις κάτω χώρες, αλλά θα πρέπει να τις προωθήσουμε. Γιατί πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλούμε για ε, επιστημονικές ε, δυνατότητες, αλλά δεν μιλούμε για τεχνολογικές δυνατότητες. Ε, πάλι επικεντρωνόμαστε στην επιστήμη. Δεν μιλώ για περισσότερα κονδύλια, αλλά περισσότερο για πιο ευφύ αξιοποίησή του. Υπάρχει μεγάλη ανισότητα, δαπανούμε τεράστια κονδύλια στις βασικέ επιστήμες, αλλά όχι στην τεχνολογία, δεν έχει νόημα. Ενώ οι άλλοι επενδύουν περισσότερες τεχνολογίε. Υπάρχει λοιπόν τέτοια αποσύνδεση πανεπιστημίων από αγορά. Θα έχουμε τα στοιχεία για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να, να χρηματοδοτούμε προγράμματα. Βλέπετε σε μια κλίμακα 1 έως 10 οι τεχνολογίες ε, ένα είναι οι βασικές επιστήμες και δέκα στην κλίμακα είναι το πρόγραμμα στην αγορά. Μέχρι την κλίμακα 4 δυστυχώς χρηματοδοτεί προγράμματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το 1 στο 4. Το 5 που είναι πρωτότυπα ε, και εργαστήρια τα φοβούνται γιατί ότι θα είναι πολύ κοντά στην αγορά. Ενώ οι Ηνωμένε χρηματοδοτούν από την κλίμακα 1 έως 8. Το ίδιο και οι ασιατικές χώρες. Χρηματοδοτούν σχέδια έως 8. Υπάρχει αποσύνδεση λοιπόν πανεπιστημίων και αγοράς. Και έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες και ε, εμπειρογνώμονες, αλλά δεν ε, τους επιτρέπουμε να φέρουν την επιστήμη πιο κοντά στην αγορά. Δεν υπάρχουν νομικά κολλήματα δεν υπάρχουν προβλήματα με τους κανονισμούς. Ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει ερευνητικά σχέδια από το επίπεδο 1 στο 8 και όχι μόνο μέχρι το 4 και θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή της βιομηχανίας σε προγράμματα πλαίσιο γιατί έχει, έχει μειωθεί ε, δραστικά η συμμετοχή της βιομηχανίας από τα προγράμματα. Έχει μειωθεί σταδιακά η, η συμμετοχή της βιομηχανίας από τα προγράμματα πλαίσιο γιατί οι βασικές τεχνολογίες ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα και για να πετύχουν χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσαρμοστούν σε βασική έρευνα. Δεν έχει νόημα για αυτού. Υπάρχει αποσύνδεση, θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Έχουμε εξαιρετικού ε, εμπειρογνώμονε, θα πρέπει να του δώσουμε πολεμοφόρητα για να δώσουν τη μάχη του. Διατομιακή προσέγγιση, το είπαμε και προηγουμένω. Έχουμε φωτονικά στη Γενική Διεύθυνση Ήψων, έχουμε τα υλικά στη Γενική Διεύθυνση Έρευνα και Καινοτομία για φωτονικά χρειαζόμαστε νέα υλικά. τι ο κατακαιρματισμός, δεν έχει νόημα. Τι νέες ε, ε, ικανότητες χρειαζόμαστε. Στην έκθεση μιλούμε για τρεις πυλώνες. Πρώτος, ε, πυλώνας τεχνολογικής ικανότητας για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας. Να στηρίξουμε τις οργανώσεις εφαρμοσμένης έρευνας. Να είμαστε υπερήφανες για αυτές, να τους δώσουμε πρόσβαση στην ε, χρηματοδότηση και την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για προγράμματα και εφαρμοσμένης ε, έρευνας. Και να μην πει κανείς ότι ένα τέτοιο προϊόν είναι κοντά στην αγορά. Νομίζω ότι εκεί έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε για να εφαρμόσουμε στο επόμενο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο μια πραγματικά διατομιακή προσέγγιση. Κύριε Τροτμάν, τρία σχόλια ε, υποβάλλατε. Αναφερθήκατε καταρχήν στους κανόνες. Στους κανόνες του παιχνιδιού στην Ευρώπη βρισκόμαστε με δεμένα χέρια. Ακόμη και αν μία χώρα θέλει να υποστηρίξει μια βασική εταιρεία σε σημαντικό κλάδο, κρόκους ε, στην Κρενόμπλη για παράδειγμα. Ακόμη και αν το επιθυμεί μια χώρα δεν μπορεί να εξασφαλίσει 50% σε χρηματοδότηση για την εταιρεία της. Γιατί θα προσκρούσει στις ε, ενστάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού παρόλο που και η εταιρεία θα συμβάλλει και θα προσφέρει πολλά εκατομμύρια. Γι' αυτό φεύγουν οι βιομηχανίες, οι επιχειρήσεις από την Ευρώπη. Δεν είναι οι ίδιοι οι του παιχνιδιού. Δεν υπάρχουν συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού. Θα είχαμε πολύ περισσότερες δαπάνε στις βιομηχανίες αν ε, διευκολύναμε τον κλάδο αυτό. Πολλοί αναφέρθηκαν στην Κίνα. Φυσικά δεν θέλουμε εμεί να αντιγράψουμε το σύστημα τη Κίνα. Έχουμε άλλε αρχέ και αξίε. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά γιατί να μην μιμηθούμε τι Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί αν οι Ηνωμένε Πολιτείε μπορούν να εντοπίσουν συγκεκριμένε εταιρείε ε, και τομεί και να προσελκύσουν τις αντίστοιχες ε, εταιρείες από την Ευρώπη για μαγνητική μνήμη για παράδειγμα ή διάφορες ε, ε, εταιρείε από την ε, Γερμανία, την BASF για παράδειγμα, για τις μπαταρίες. Γιατί να μην κάνουμε κάτι τέτοιο κι εμεί, γιατί να μην ανταγωνιστούμε κι εμεί στι Ηνωμένε Πολιτείε, Χρειαζόμαστε ευφιέστερου κανόνες, ε, ρυθμίσει, διατάξει και ευφιέστερη αξιοποίηση των κονδυλίων. Στις 26 Σεπτεμβρίου θα μιλήσουμε για τι ρήτρε αντιστοίχηση, ώστε να δημιουργήσουμε ένα παραλληλισμό και στην Ευρώπη των κινήτρων που δίνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Να έχουμε και εμεί εφάμιλα κίνητρα και ανάψματα. Θα το συζητήσουμε αυτό το Σεπτέμβριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε ολοκληρωμένη προσέγγιση να περάσουμε αυτή την κοιλάδα του θανάτου να δώσουμε έμφαση σε τεχνολογικές υποδομές, σε τεχνολογικές επενδύσεις και κάποιες ε, πιλωτικές γραμμές και δυνατότητα της βιομηχανίας για πρότυπα μοντέλα. Χρειάζεται αυτό για τις βιομηχανίες. Θα πρέπει να κατασκευάστε τα πρωτότυπα για να μεγαλώσει το μερίδιό τους στις μεγάλες αγορές. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τι βιομηχανίε μας σε αυτή την προσπάθεια. Θα πρέπει λοιπόν να χρηματοδοτήσουμε και πιλωτικά προγράμματα. Κύριε Λάμπερτ, είπατε ότι στο μέλλον το μεγαλύτερο τμήμα της χρηματοδότησης θα είναι ιδιωτικό. Συμφωνώ, θα πρέπει να επιτρέψουμε και να διευκολύνουμε τη βιομηχανία να δαπανίσει αυτά τα κονδύλια. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στις κοινέ τεχνολογικές πληροφο... Ε, πρωτοβουλίες της Γενικής Διάθεσης ΣΥΜΣΟ. Πέρυσι είχαμε 400 εκατομμύρια που έμειναν ανεκμετάλλευτα γιατί δεν μπόρεσε η βιομηχανία να υποβάλει ένα πρόγραμμα υπό αποδεκτούς όρους και έτσι τα, τα κράτη-μέλη δεν μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τέτοια πρόγραμμα με αποδεκτούς όρους μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα και μια, μικρή αλλαγή στον κανονισμό, ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να συγχρηματοδοτήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συνεπενδύσουν, αντί να βάζουν όλα τα χρήματα σε ένα κοινό πουλ. Μια τέτοια μικρή αλλαγή θα προκαλούσε τεράστιες επενδύσεις από τη βιομηχανία. Σε ό,τι αφορά τη Γενική Διεύθυνση ύΜΣΟ, συνεργάστηκα με πολλές βιομηχανίε ηλεκτρονικών και είχαμε βιομηχανικά σχέδια ύψους ενός δισεκατομμύριου ευρώ με 50% επενδύσεις από τη βιομηχανία. Και με μία μικρή αλλαγή τον κανονισμό στα JTI, στους κανόνες για τις ε, κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες, θα αρκούσε για να ε, συνεπενδύσουν 500 εκατομμύρια και το καταφέραμε μέσα σε λίγους μήνες. Πήγαμε στην ε, αρμόδια επίτροπο, την Έλλη Κρούς, και τι είπαμε 400 εκατομμύρια έμειναν αχρησιμοποιητά πέρυσι επειδή ούτε η βιομηχανία ούτε τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να συγχρηματοδοτήσουμε του τους αποδεκτούς Κοιτάξτε, μια μικρή αλλαγή των κανόνων, τι κέρδο θα έχουμε. Συμφωνώ μαζί σα ότι χρειαζόμαστε ιδιωτικέ εμπεδίσει, θα πρέπει να τι ε, ενθαρρύνουμε και όχι να τι ε, παρακολύσουμε. Επίση κινητοποίηση γύρω από μεγαλεπίβολα σχέδια. Συμφωνώ και σε αυτό Ιδιαίτερα στις βασικές τεχνολογίες χρειαζόμαστε μεγάλες ε, επιχειρήσεις και ε, ε, δυναμικό κατασκευής παγκόσμιας κλίμακας. Και αυτό το χάνουμε εξαιτία των εσωτερικών κανόνων ανταγωνισμού. Ο πρόεδρος είναι Γερμανός, σας θα το παράδειγμα της, Γεωργίας, της Γερμανίας. Συγγνώμη. Στη Δρέσδη είχαμε ε, σημαντική εταιρεία στην κατασκευή μικροελεκτρονικών. με πρωταγωνιστικό ρόλο παγκοσμίω στη μικροελεκτρονική. Αν δεν κάνω λάθος, οι επιδοτήσεις από την κεντρική κυβέρνηση ήταν το 28%. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, κύριε Πρόεδρε. Πριν από μία οκταετία. Πέρυσι, η AMD ε, διεκδικήθηκε από άλλον επενδυτή και είπαν ότι χρειαζόταν μια αναβαθμισμένη ικανότητα. Δεν ήταν ανταγωνιστικές οι τιμές. Οι επενδυτές ήταν πρόθυμοι να προσφέρουν δισεκατομμύρια ευρώ και το μόνο που ζήτησαν ήταν η ίδια επιδότηση από τη γερμανική κυβέρνηση, την Ομοσπονδιακή και τους ε, ενδιαφέρομενους. Ήταν θετική απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης. Γιατί πραγματικά ήταν λειτουργική μονάδα, υπήρχαν υποδομές, αλλά υπήρξε η αντίδραση από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού που δεν έδωσε το πράσινο φως για το 28%. Ανώτατο για αυτούς όρικτο το 15%. Αποτέλεσμα έφυγε από το εργοστάσιο και πήγε στι Ηνωμένε Πολιτείε. 2.000 θέσει απασχόληση δημιουργήθηκαν στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει εκεί ένα ε, εργοστάσιο προηγμένη τεχνολογία, ενώ το εργοστάσιο τη Δρέσδη ε, ε, το μέλλον του πια έχει υπονομευθεί εξαιτία των ε, κανόνων ε, ανταγωνισμού που μπλοκάρει τη δράση των κρατών μελών. Και η συνολική επιδότηση ήταν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Η απόδοση όμως στην Ευρώπη από το συνολικό τζίρο αυτού του εργοστασίου και είχαμε την Ιντελ και στην Ιρλανδία είχαμε εταιρείε, είχαμε την αντίστοιχη της Γερμανίας. Η ετήσια απόδοση για την οικονομία είναι πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Έχουμε όλα τα στοιχεία και θα μπορούσαμε να σας τα μεταφέρουμε. Μέσα σε δύο χρόνια θα κατάφερε να αποσβέσει αυτή την επιδότηση η γερμανική κυβέρνηση. Ταχύτατα λοιπόν και παρόλα αυτά δεν δόθηκε το πράσινο φως. Και έτσι υπονομεύθηκε ανεπανόρθωτα η μικροηλεκτρονική στη Γερμανία εξαιτία αυτή τη ε, διαφυγή και τη άρνηση τη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η βιομηχανία θέλει να επενδύσει και μάλιστα είναι πρόθυμη να επενδύσει τεράστια κονδύλια. Και μάλιστα στην ομάδα εμπειρογνωμών υψηλού επίπεδου είχαμε πολλές συναντήσεις με εκπροσώπους βιομηχανιών και μας εξέφρασαν την επιθυμία αυτή της επένδυσης και μάλιστα το παράδειγμα αυτό της απώλειας του εργοστασίου στη Δρέσδη και τη διαφυγής προς την ΕΠΑ ήταν μάθημα για τη Γερμανία. Φυσικά μπορούμε να σας ε, μοιράσουμε αντίγραφο της έκθεσης και της παρουσίασης. Κινητοποίηση του κεφαλαίου. Φωτοβολταϊκά δεν είχαν τις απαραίτητες ε, αποδόσεις. Δυστυχώς το όλο ζήτημα των φωτοβολταϊκών ήταν παταγώδης αποτυχία. Το μεγαλύτερο ερευνητικό Ινστιτούτο στην ε, Γερμανία είναι το Ινστιτούτο Φωτοβολταϊκών στη, Φρα, στη Φράιμπουργκ. Χίλια άτομα προσωπικό. Τεράστιο Ινστιτούτο. Οι περισσότερες επιδοτήσεις στον κόσμο για τα φωτοβολταϊκά δίνονται στην Γερμανία. Και μόνο ένα εργοστάσιο έχει μείνει, που δεν είναι ούτε καν μέσα στα 10 καλύτερα ή δεν θα, είναι, δεν θα παραμείνει του χρόνου. Κάτι πάει στραβά λοιπόν. Έχουμε τη μεγαλύτερη αγορά φωτοβολταϊκών στον κόσμο, τι περισσότερε επιδοτήσει, τη μεγαλύτερη επένδυση στη, στην έρευνα και ένα, μια τεράστια τρύπα στο κέντρο γιατί δεν δίνουμε τα απαραίτητα κίνητρα. Κάτι πάει στραβά λοιπόν. Σίγουρα για τα φωτοβολταϊκά δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αν πρέπει να θέσω μια ευρύτερη προσέγγιση, φυσικά δεν μιλούμε μόνο για χρήματα εδώ. Θέλουμε η πνευματική ιδιοκτησία να αξιοποιηθεί πρώτα απ' όλα στην Ευρώπη. Και θέλουμε να αξιοποιήσουμε στην ευρωπαϊκή πολιτική την πνευματική ιδιοκτησία. Γιατί όχι. Δεν υπάρχει λόγος να μην γίνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα πολύ σύντομα θα πρέπει να τεθεί αυτή η ρήτρα σε όλες τις διαπραγματεύσεις συμβάσεων. Κάνει; δεν θέλουν να υπογράψουν, εντάξει. Η Ωστραμ, η Infineum, η Philips, μεγάλες εταιρείες που συμμετέχουν σε επιχείρημιση στις Ηνωμένε Πολιτείες και σε προγράμματα που χρηματοδοτούν οι Ηνωμένε Πολιτείες από το Υπουργείο Ενέργειας και τα αποτελέσματα της έρευνας που κάνουν οι εταιρείες αυτές τα ε, χρησιμοποιούν στις Ηνωμένε Πολιτείες. Μεγάλες επιχειρήσεις ακολουθούν τους αμερικανικούς κανόνες και εμείς εδώ δεν κάνουμε τίποτα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε το 2014 για να κάνουμε κάτι. Θα πρέπει να υπάρξει μια έκκληση και από το Κοινοβούλιο. Πρέπει να δούμε την κατάσταση με διαφορετικό τρόπο το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και θέμα αριθμίσεων. Τώρα για τα σχόλια που έκανε η συνάδελφος από την Ουγγαρία. Το θέμα δεν είναι περισσότερα χρήματα μόνο, είναι χρήματα τα οποία δαπανώνται σωστά. Το παράδειγμα που σας έδωσα για τα χρήματα που περίσσεψαν από πέρυσι είναι ένα από τα παραδείγματα. Μέσω μιας διαφορετικής μικρής ρύθμισης στους νόμους μπορεί να κερδίσει κανείς πάρα πολύ. Και το λέμε αυτό στην έρευνα. Συνεπώς, μπορούμε να έχουμε κάποιους κανόνες οι οποίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να παίρνουν μέρος σε όλες αυτές τις μορφές χρηματοδότησης. Και φυσικά θα κάνουμε και μία παρουσίαση και προς το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, μετά από το δικό σας αίτημα βέβαια πάντα. Περνάω τώρα στα σχόλια την οποία έκανε η κυρία Βαν σχετικά με τα κρατημέλη. Φυσικά, τρεις υπουργοί υπέγραψαν ε, την κοινή επιστολή. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία έχουμε δώσει, στα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε 14 ομάδες εργασίας με τους καλύτερους ηγέτες της αγοράς. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν. Συμφωνώ και με τα στοιχεία που έγιναν ε, σχετικά με τα νέα εργοστάσια σε πολλές περιοχές όπως επίσης και σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Κορέα. Μπορούμε να σας δώσουμε επιμέρους στοιχεία αν χρειάζεστε. Και για τα τελευταία σχόλια, για το πώς θα μπορέσουν οι περιφέρειες να συνδοθούν με τις προσπάθειες αυτές, εμείς ζητήσαμε να είναι δυνατό να συνδυάσει χρηματοδοτήσεις κανείς από διαφορετικές πηγές για ένα πρόγραμμα μεμονωμένο. Και στα πλαίσια των συζητήσεων με τον Επίτροπο Χάν, νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα και τα ΚΕΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να συνδυάσουμε πρωτοβουλίες με τα διαρθρωτικά ταμεία και με κάποια προγράμματα πλαίσιο. Νομίζω ότι τότε μπορούμε πράγματι να προχωρήσουμε. Πρέπει να υπάρξουν ορισμένες τεχνολογίες, ορισμένοι τομείς που θα επιλεγούν από τις περιφέρειες να συνδεθούν με κάποιες πρωτοβουλίες έρευνας, ερευνητικές και έτσι τα πράγματα σίγουρα μπορεί να επιταχυνθούν. Στην παρούσα φάση καταλαβαίνετε ότι είναι τρομερές δυσκολίες να μπορέσει να συνδυάσει κανείς κανόνες για τις δαπάνες με διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, γιατί οι ρυθμίσεις και οι κανονισμοί χρηματοδότησης είναι εντελώς διαφορετικοί. Λοιπόν το θέμα, επαναλαμβάνω, δεν είναι να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα, αλλά να μπορέσουμε τα χρήματα αυτά να τα συνδυάσουμε σωστά. Δυστυχώς όταν προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό στο παρελθόν και με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας υπήρξαν πάρα πολύ σημαντικοί δισταγμοί. Αλλά παρόλα αυτά οι περιφέρειες, οι πόλεις, οι τοπικές αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο και αυτό μπορεί να προκαλεί και επιπλέον δυσκολίες μερικές φορές. Νομίζω ότι συμφωνώ και με τα περισσότερα σχόλια τα οποία κάνατε για τις, για τις επιπτώσεις σε διάφορες τομείς. Ελπίζω να κάλυψα, εν πάση περιπτώσει, κάποια από τα σχόλιά σας. Μην διστάσετε να έλθετε σε επαφή μαζί μου αν θέλετε και στο μέλλον κάποιες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ θερμά. Να σας ανακοινώσω ότι ε, αύριο θα λάβουν όλοι οι συνάδελφοι την παρουσίαση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ε, κλείνω τη σημερινή συνεδρίαση. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί.